Um, Συνάδελφοι, καλησπέρα. Ίσως να υπάρξει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα με τον Πρόεδρο, ο οποίος καθυστέρησε ένα δεκάλεπτο και ζητώ συγγνώμη. Είναι μία από αυτές τις ημέρες, ξέρετε. Το έκανα δύο φορές σήμερα, συνήθιστο. Ζητώ συγγνώμη. Και δεν έχουμε και πολλούς συναδέλφους παρόντες. Κύριε Μπόνη, εσείς μας στηρίζετε αν μπορώ να δώσω ένα βραβείο, ένα παράσημο, θα δημιουργήσω παράσημο για την Επιτροπή μας, θα ο πρώτος για την απονομή του. Δεν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά θα το πάρω το παράσημο. Και στο προσωπικό θα δώσω κάποια παράσημα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ίσως να έχουμε πρόβλημα, διότι ξεκινάμε κανονικά στις 2. Κανονικά άλλες φορές ξεκινάμε στις 3 και σήμερα στις 2. Ζητώ συγγνώμη από όλους, ήταν ασυνήθιστη ημέρα Είχαμε ψηφοφορίες, συναντήσεις κλπ. Συγγνώμη σε όλους και κυρίως στους φιλοξενούμενους που ήρθαν. Μεταδίδεται και στο διαδίκτυο η συνεδρίαση και πολλοί θα παρακολουθούν. Είναι πέμπτη και πολλοί έχουν κανονίσει ε, να ταξιδέψουν και πολλοί έχουν κανονίσει να παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε. Κύριε Μπόνη, θα αντέξατε, θα είσαστε ικανοποιημένο να μείνετε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια τη σα. Α, για το μεγαλύτερο τμήμα τη. Αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε και άλλο πλήρε μέλο εδώ, ω επισκέπτη. Μόνο ένα μέλο έχουμε. Ωραία. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα συνεχίσουμε. Δεν είχα άλλη φορά τόσο ολιγάριθμη παρουσία. Είναι διαθετικό θέμα, ξέρετε. Έτσι που ε, εξελίχθηκε η μέρα. Είχαμε ψήφο για την PNR, για το PNR και λοιπά, ήρθαν πολλοί για την ψηφοφορία και έφυγαν. Δομικές αλλαγές είχαμε σήμερα τέλος πάντων. Ας ξεκινήσουμε. Σημείο 7, 8 και 9. Η αξιολόγηση του οργανωμένου εγκλήματος στο διαδίκτυο, παρουσίαση της εκθέσεως της 30 Σεπτεμβρίου από τον υποδιευθυντή του υπεύθυνο για τις επιχειρήσεις της Europol, τον κύριο Γκέμερτ, θα δούμε και ποιες είναι οι προκλήσεις όσον αφορά το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και πώς μπορούμε να επιβάλλουμε τον νόμο, αν μπορούμε πραγματικά να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Μετά έχουμε τη μελέτη για την κυβερνοασφάλεια, πέρα από τις απειλές, ποια ήθη η ανταπόκριση στις απειλές ε, σε σχέση με πολιτικές. Παρουσίαση από τον Dr. Nicole Van και την κυρία Έων ε, από την RAND Ευρώπη, το γραφείο της, ε, του Cambridge. Το πρώτο κομμάτι της συζητήσεως θα δώσουμε στον κύριο Βαν Γκέμερτ, στον υποδιευθυντή της Europol, για να μας παρουσιάσει την αξιολόγηση για τις επιλές στο διαδίκτυο για 10 με 15 λεπτά, ο κύριος Βαν Γκέμερτ. Και μετά πάμε στην καθηγήτη του πολιτικών επιστημών κλπ. Θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία που προβλέπεται στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κ. Βαγκεμέρτ. Ευχαριστώ που με καλέσατε να σας παρουσιάσω το θέμα αυτό, το ΙΟΚΤΑ. Θα ξεκινήσω λοιπόν από άλλο θέμα που πριν μια εβδομάδα ολοκληρώσατε. Κανονισμός της Europol. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και να συγχαρώ τον κύριο Δεμέρα για την δουλειά που έκανε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το θέμα ο κανονισμός της Europol, περιπλοκότατο θέμα, είχε πολλές συνέπειες, χρειάστηκε και χρόνο. Λόγω της δικής σας θέσεως και της Λουξεμβουριανής Προεδρίας υπήρξαμε επιτυχείς, ολοκληρώθηκαν συζητήσεις. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων νομικών πλαισίων από τη μια και της διαφυλάξεως των πολιτικών ελευθεριών και των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών μας από την άλλη δεν θα ήταν καλό να μην εκφράσω την ευγνωμοσύνη του υπηρεσίας μου, της Europol, ε, για αυτά που καταφέρατε. Να σας δώσω λοιπόν μια επισκόπηση των απειλών στον κυβερνοχώρο, όπως τα βλέπει η Europol, και δράτω με της ευκαιρίας να σας δώσω κάποια εικόνα όσον αφορά τις σημαντικές προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ο διευθυντής μου ήταν εδώ τον περασμένο μήνα, αναφέρθηκε στην τρομοκρατία, μετά συζητήθηκε η κρίση της μετανάστευσης, εξωτερικές σχέσεις κλπ. Θα μιλήσουμε για το κυβερνοχώρο, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, επιχειρησιακό θέμα και πάντα μας αρέσει να συζητούμε μαζί σας με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, να σας πω για το κέντρο, το ευρωπαϊκό, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 στην Ευρωπόλ για να ενισχύσουμε την ανταπόκριση Ευρωπαϊκή Ένωση στα εγκλήματα του κυβερνοχώρου. Και ένα από τα βασικά στοιχεία αναφέρθηκαν και σε άλλες εκθέσεις. Ε, δόθηκε εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασιστήκαμε στην τεχνογνωσία μας και εφαρμόσαμε τη σωστή προσέγγιση για να καταπολεμήσουμε το ηλεκτρονικό έγκλημα. Η πρωτίστως έχει καθήκον να είναι μια βάση ανταλλαγής πληροφοριών που βασίζεται και σε δίκτυο με πάνω από 200 αξιωματικούς ε, συνδέσμους, 28 κράτη-μέλη και 25 μη κράτη-μέλη. Έχουμε και κέντρο συντονισμού. Εκεί οργανώνονται μεγάλες αστυνομικέ επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς εταίρους, όπως Interpol και με τις ΙΠΑ Κολομβία, Νορβηγία και άλλες χώρες. Να πω ότι λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο πολύ ισχυρό για την προστασία των δεδομένων και θα βελτιωθεί περαιτέρω το πλαίσιο αυτό, θα ισχυροποιηθεί έχουμε ευστιαστεί σε τρεις τομείς του ηλεκτρονικού ε, εγκλήματος. Πληρωμές, απάτες όσον αφορά στις, ε, στις συναλλαγές στο διαδίκτυο, κλοπή ταυτότητας, ε, κλοπή στοιχείων πιστοτικής κάρτας κλπ. Και μετά εκμετάλλευση των παιδιών, σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που απειλούν τις διάφορες υποδομές πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε το 2015 ήδη κάνουμε, κάνει πάνω από 100 επιχειρήσεις πολύ σημαντικές. Με εφταμελές προσωπικό. Ο πιο καινοτόμος τρόπος ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μα όσον αφορά τους τζιχαντιστές, Λοιπόν, και τα κράτη-μέλη καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να μοιραζόμαστε πληροφορίες εκτός σύνορων, πέρα από τα σύνορα. Ξεπερνάμε τα όρια της συνήθους ε, ε, συνεργασίας ε, να αντιμετωπίσουμε στο θέμα, το θέμα αυτό του προβλήματος των τζιχαντιστών στον, στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Έχουμε αξιωματικούς συνδέσμους από 7 κράτη-μέλη που συμμετέχουν και από 4 χώρες μη μέλη και, και τονίζουμε προτεραιότητες όσον αφορά τους στόχους και τις έρευνες που πρέπει να γίνουν και ο τρόπος δεν τα εξετάζουμε από εθνική σκοπιά, αλλά υπερεθνική τα προβλήματα. Και ούτω τρόπο αποφασίζουμε ποιο είναι ο καλύτερο τόπο αντιμετωπίσεω του προβλήματο. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε συνεργασία και με άλλου φορεί. Και τα κράτη-μέλη συνεργάζονται και τα μη κράτη-μέλη. Έχουμε νέε προσεγγίσεις λοιπόν που ακολουθούμε. Και Τώρα όσον αφορά το τοπίο του ηλεκτρονικού εγκλήματος το 2015 κινήθηκε, έχουμε το IOCTA που είναι στατηγική αξιολόγηση που κάνουμε για το οργανωμένο έγκλημα στον κυβερνοχώρο και το 2015 ε, ε, βλέπουμε την ε, οπτική γωνία της επιβολής του νόμου και διαφέρει από άλλες αξιολογήσεις του ιδιωτικού τομέα. Στόχος του εγγράφου. Να δούμε το μέλλον. Στατική επισκόπηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Θέλουμε να ενημερώνουμε εκείνους που θεσπίζουν νομοθεσία, να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις, για τα προβλήματα, για τις επιτυχίες. Βασιζόμαστε σε συνδρομή 28 μελών, αλλά από τον ιδιωτικό τομέα, τον οικονομικό τομέα, τα πανεπιστήμια που μας συνδράμουν. Ποια είναι τα βασικά πορίσματα της μελέτης. Το ηλεκτρονικό έγκλημα δεν αποτελεί μυστικό ότι γίνεται πιο επιθετικό και οδηγούμεθα σε μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις. Είναι καινούριο αυτό σαν φαινόμενο και αναμειγνύεται όλο και περισσότερο απειλές, εκβιασμοί προς άτομα, προς εταιρείες και ασκούνται μέσω του κυβερνοχώρου, ανοιχτές, ανοιχτοί εκβιασμοί ε, και έτσι διαπράτεται ένα, ένα κομμάτι του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Λόγω της διαθεσιμότητας της δυνατότητας ε, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και κάποιοι που αρχικά είναι αδέξεις αυτό μαθαίνουν και τελικά γίνονται πιο επιθετικοί και αυξάνουν τον όγκο των επιθέσεων. Λοιπόν, ε, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο όσον αφορά την κρυπτογράφηση. και Δύο τρίτα των κρατών μελών κάνουν έρευνα όσον αφορά το θέμα αυτό για τους εκβιασμούς κλπ. Είχαμε, είχαμε κάνει λοιπόν μια επισκόπηση και μια έρευνα πέρσι. Α, και ήταν και η χρήση σε κακού λογισμικού malware που απειλεί εκείνον που είναι θύμα και εκβιάζουν ζητώντας χρήματα. Λοιπόν, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα φαινόμενα της χρήσης malware έχουμε σε επαφή με ιδιωτικούς εταίρους, προσπαθούμε να εντοπίσουμε και τα θύματα και να βοηθήσουμε τα θύματα και να τους δώσουμε εργαλεία για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση αρχείων, ούτως ώστε να είναι ασφαλή. Και υπάρχει αυτό το malware λοιπόν που τελικά μπλοκάρει τον υπολογιστή σου και αν δεν δώσεις χρήματα δεν, ε, δεν ξαναλειτουργεί. Και βρήκαμε όμως έναν τρόπο να ξεκλειδώνουμε αυτό το παράνομο κλείδωμα. Επίσης ε, γίνονται και επιθέσεις κατά του online banking και γίνονται όλο και πιο περίκλοκες επιθέσεις. Οι τεχνολογίες εξελίξεις τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό ε, έγκλημα, ε, η αποκάλυψη διαφόρων στοιχείων κλπ. κλπ. και νέο λογισμικό που συνεχώς αναπτύσσεται. Και γίνεται όλο και πιο δύσκολο να καλυφθούν τυχόν κενά στο λογισμικό. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν δοκιμασμένες μεθόδους επίθεσης και στις αδυναμίες των συστημάτων. Άρα εκεί τα κενά και τις αδυναμίες μπορούμε να τα, να τα ε, καλύψουμε. Τώρα εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες τα συστήματα κρυπτογράφησης και τα ε, υγικά συστήματα, τα αντιβάρους. Το 2015 στην Ευρώπη πάνω από 3-4 των ερευνών που κάναμε αφορούσαν τη μορφή κάποιας κρυπτογράφησης για την προστασία των στοιχείων και των επικοινωνιών και σε πρόσφατο μεγάλο πρόβλημα σε επιχείρηση που κάναμε, το Jet Mozart, είδαμε ότι 62% των μηνυμάτων που είχαν ανταλλαχθεί από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και αυτοί χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένα συστήματα, λογισμικό κρυπτογράφησης και έτσι δεν μπορούσαμε να ε, δούμε ακριβώς τα μηνύματα που ανταλλάσσουν. Και δεν μπορούσαμε να αποκτήσουμε και στοιχεία Άρα τα παραδοσιακά εργαλεία της αστυνομίας για να παρακολουθούμε τους εγκληματίες ε, γίνονται λιγότερα αποτελεσματικά όπως οι παρακολουθήσεις τηλεφωνημάτων. Η αστυνομία λοιπόν δεν μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματική. Το ίδιο ισχύει όταν θέλουμε να κάνουμε συλλήψεις και όταν πιάσουμε τον σερβερ, ε, κατάσχουμε τον, ε, τον, τον σερβερ του εγκληματία, δεν είναι εύκολο να αποκρυπτογραφήσουμε τα στοιχεία που εμπεριέχεται για να έχουμε στοιχεία να κινηθούμε εναντίον τους, γιατί είναι κρυπτογραφημένα και αυτό είναι απογοητευτικό για μας. Και κάτι άλλο. Η Europol εκ, ποτέ δεν ζητούσε ε, διάφορα, τα διάφορα λογισμικά να τους δίνουν δυνατότητες δίδυσης για να παρακολουθούν τους ιδιώτες στις συναλλαγές, τα λεγόμενα backdoors. Υπάρχει σημαντική διάκριση να κάνουμε μεταξύ της κοινότητας της ευρωπαϊκής επιβολής του νόμου και των μυστικών υπηρεσιών και μπορεί να έχουμε και διαφορετικές απόψεις αφορείς. Στη Europol γνωρίζουμε ότι χωρίς ισχυρή κρυπτογράφηση δεν λειτουργούσε τώρα το διαδίκτυο, ούτε στο μέλλον, ιδιαίτερα στο μέλλον. Αντιθέτως ζητάμε να υπάρξει νομοθεσία που θα δίνει ισορροπημένες εξουσίες στην κοινότητα επιβολής του νόμου, τόσο ώστε να συνεχίσει να συμβάλλει στην, στο σύστημα καταπολέμησης του εγκλήματος και να γίνονται οι έρευνες και η δίωξη του εγκλήματος. Έτσι θα εξασφαλίζονται και τα δικαιώματα των θυμάτων και των πολιτών, θα προστατεύονται. Υπάρχουν κάποια αναλλακτικά μέτρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να λάβει για να πετύχει σωστή ισορροπία και να μειώσει τα προβλήματα χωρίς να υπονομεύει την τεχνολογία διότι αυτό θα ήταν η περίπτωση των backdoors, δηλαδή διεξόδων για να μπορούν να διεισδύει η αστυνομία και να ε, αναλύει τα στοιχεία που είναι κρυπτογραφημένα. Τούτων λεχθέντων λοιπόν στρεφόμαστε προς την ΑΙΟΚΤΑ χρησιμοποιούν το bitcoin για να δούμε τα ηλεκτρονικά νομίσματα. Ε, όχι μόνο για εκβιασμό αλλά και για πολλά άλλα δικήματα πρέπει να εφαρμόσουμε τον ίδιο κανονισμό κατά του ξεπλήματος χρήματο και εδώ, με το ηλεκτρονικό χρήμα, και το εικονικό χρήμα, όπως κάνουμε και στον πραγματικό χρηματοστατικό τομέα. Ε, θα πρέπει να αναλαμβάνονται ιδέουσες ευθύνε έναντι των πελατών. Πριν ολοκληρώσω κάποια πορίσματα, το 2014 ήταν το έτος παραβιάσεως των στοιχείων, η κοινωνική μηχανική ε, παίζει μεγάλο ρόλο και στον τομέα των απατών και για την, κατά, για την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών έχουμε μεγάλη αύξηση λόγω της ζωντανής μετάδοσης ε, εικόνων από την παιδική πορνογραφία. Ε, και επίσης υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα για τους νέους πολίτες αυτή η παραγωγή αυτών των, του πορνογραφικού υλικού που μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Λοιπόν, κάποιες συστάσεις που από την έκθεση. Για να είμαστε αποτελεσματικοί για τη μετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Οι νομοθέτες πρέπει να μας δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία, παιδεία, κατάρτιση, για να μπορούμε να κάνουμε τις αναγκαίες έρευνες και να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση της κωδικοποίησης των στοιχείων και, και α, ε, της Χρειάζεται λοιπόν συνδρομή όλων. Πρέπει να εστιαστούμε στην πρόληψη, στην ευαισθητοποίηση, στην εκπαίδευση, δημιουργία δυναμικού εντός αστυνομικών αρχών κλπ. Πρέπει να προστατεύουμε τα θύματα, να τα σώζουμε. Μέσω της ταυτότητας του θύματος που να διαπιστώνεται. Χρειάζεται εναρμόνιση τη νομοθεσία για αυτό το σκοπό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται μέτρα για να μειωθούν τα αποτελέσματα τη κρυπτογράφηση, να έχουμε ρεαλιστική νομοθεσία για τα εικονικά νομίσματα και να υπάρχει νομικό πλαίσιο ευρωπαϊκό για την διατήρηση των στοιχείων. Τι ο τρόπο μπορούμε να πετύχουμε σωστή ισορροπία μεταξύ ιδιωτική ζωή και επιβολή του νόμου. Απαιτείται πολιτικό θάρρο, υψηλό αίσθημα ευθύνη για να επιτευχθεί η συνένεση του λαού που απαιτείται μετά τα Snowden links. leaks. Λοιπόν, με την εξέλιξη του χρόνου εξελίσσεται και το έγκλημα. Χρειάζεται προστασία ο πολίτης. Και εμείς, σαν Ιωπόλ, με τα χαράς να βοηθήσουμε να επιτευχθούν οι στόχοι των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Ευχαριστώ. Um, Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη παρουσίαση θα ακούσουμε την ε, παρουσίαση ε, από το Πανεπιστήμιο ε, και από το Κέντρο για την μελέτη σχετικά με τις συγκρούσεις, την ελευθερία και την ασφάλεια. Great. Thank you. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Εξ ονόματος του συναδέλφου μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας και να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης που κάναμε ε, για το ε, ηλεκτρονικό έγκλημα. Ποια είναι τα προβλήματα. Ε, Πρέπει να τα εντοπίσουμε πρώτα και να τσιάσουμε στα θέματα της κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ε, στα διάφορα λογισμικά και τα λεγόμενα εικονικά νομίσματα, κρυπτονομίσματα όπως είναι το bitcoin. Ε, είναι τριπλό το πλαίσιο. Από τη μια θέλουμε να εστιάσουμε ε, στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστήσει αυτό το τομέα ένας από τους τρεις βασικούς που την ανησυχούν στο θεματολόγιο για την ασφάλεια για το 2015. Από την άλλη, ε, ακούμε όλο και περισσότερο ότι υπάρχουν παραβιάσεις δεδομένων, hackers, όπως είπε και ο κύριος Φανχέμερτ, το 2015 ήταν ε, η χρονιά παραβιάσεων δεδομένων. Ε, hacks ε, και από malware, από κακό βουλολογισμικό. Ε, επίσης, το τελευταίο πλαίσιο είναι οι αντικρουόμενες εκτιάσεις και ισχυρισμοί ε, και ε, για το κατά πόσο χρησιμοποιούν αθέμητες μεθόδους οι αρχές τήρησης και επιβολής του νόμου και της τάξης. Και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καμιά φορά και ε, στην Ευρώπη, ότι οι υπηρεσίες κινδυνεύουν με όλους αυτές τις κρυπτογραφήσεις και τα εικονικά νομίσματα να κατρακυλήσουν σε ένα σκοτεινό δίκτυο με έκτακτες ε, ε, ρυθμίσεις για κρυπτογράφηση ε, με διάφορους τρόπους που χρησιμοποιούμε και ήδη στην καθημερινή δουλειά. Βλέπουμε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί φαίνονται να αναδύονται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη με τα μέτρα που παίρνει η γαλλική κυβέρνηση μετά τη 13η Νοεμβρίου και το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι. Άρα λοιπόν θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ποια είναι τα κύρια ευρήματά μας. Γίνεται μια συζήτηση και δημόσια και τεχνική για τα τεχνολογικά και τα τεχνικά μέσα που έχουμε για να καταπολεμήσουμε το ηλεκτρονικό έγκλημα. Τι έδειξε όμως η μελέτη, ότι τα θέματα σχετίζονται πιο πολύ με την πολιτική και με τον νόμο, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, οι τεχνολογικές δυνατότητες υπάρχουν, αλλά πώς γίνεται όλα αυτά να είναι σύνομα. Έτσι θα πρέπει να μπορεί κανείς να δρά και στη συνέχεια να διώκει και το ε, έγκλημα και το ηλεκτρονικό. Άρα λοιπόν ε, καταλήξαμε στα εξή αποτελέσματα. Τι κατέδειξε η έρευνα σχέση ε, με το σενάριο ότι θα διολυστήσει στο σκοτεινό διαδίκτυο ε, η αστυνομία ή οι αρχές. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει τεχνολογία, αλλά δεν σημαίνει ότι τέτοια ε, ακραία μέτρα όπως είναι η έκτακτη πρόσβαση θα υιοθετηθούν ή θα εξεταστούν. Ακούσαμε από τις συνεντεύξεις που κάναμε στη Europol και στη Eurojust ότι οι ανακρίσεις εδώ έχουν να κάνουν κυρίως με τεχνικές δεξιότητες, τις οποίες πάντα δεν διαθέτουν οι ίδιοι. Ούτε οι ιδιοκτικές αρχές των κρατών μελών. Ε, υπάρχει ε, τώρα μια κούρσα ε, όπλων κλέφτες και αστυνόμους παίζουμε στο ε, διαδίκτυο ε, όχι. Καμιά φορά είναι χειραγώγηση ε, και το χρησιμοποιούν για να αυξηθούν οι εντολές, ε, το πεδίο δηλαδή εφαρμογής ορισμένων δράσεων ή τα οικονομικά. Στην συντριπτική πλειονότητα το ηλεκτρονικό έγκλημα χρησιμοποιεί κάποιες δυνατότητες και κάποια ευάλωτα σημεία που υπάρχουν εδώ και κενό και, και καιρό στο διαδίκτυο. Έχουν να κάνουν με ανθρώπινους παράγοντες και ε, με μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και λιγότερο με τα τεχνικά. Ε, η έκτακτη τώρα και εξαιρετική πρόσβαση στην κρυπτογράφηση ή ε, κάποια απαγόρευση ή διάλυση κάποιων σελίδων ή δυνατοτήτων, αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Οι κλίδες κρυπτογράφησης ε, και στις έκτακτες ε, περιστάσεις ε, περιπλέκει τα πράγματα, φέρνουν ένα πλέον επίπεδο δυσκολίας. Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες να εντοπιστεί το εγκληματικό πεδίο στο ηλεκτρονικό έγκλημα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Εμείς δεν έχουμε βρει ε, καμένα ε, ορισμό για το ηλεκτρονικό έγκλημα και την ηλεκτρονική ασφάλεια στο κυφαινοφόρο για την, ε, τον πόλεμο. Δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση ούτε ενιαία μέτρα. Όσοι λοιπόν θεωρούν ότι το διαδίκτυο γίνεται ένας χώρος εγκλήματος είναι μάλλον αυθαίρετοι στις ε, τοποθετήσεις και στις ερμηνείες τους και δεν τεκμηριώνουν τόσο λέγουν. Στη συνέχεια, ε, ε, τα ευρήματα που έχουν να κάνουν με τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Δεν, μάλλον το ίδιο κοινό πρόβλημα. Δεν υπάρχει νέος ορισμός για το τι εστί έγκλημα στον χώρο. Επιπλέον, και αυτό θα το βρείτε σε πολλές μελέτες για την Επιτροπή σας, τα όρια μεταξύ κυβερ... Ε, ασφάλειας και κυβερνοεγκλήματος ε, είναι συγκεχημένα. Δηλαδή κάτι που ε, θα πατάξει το ηλεκτρονικό έγκλημα μπορεί να πατάξει και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυξάνονται και οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Europol, του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλήματος και του JCAT. Άρα υπάρχει μεγάλη επικάλυψη και μεγάλη σύγχυση σε αυτό το χώρο. Τι είναι ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τι είναι έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Η JCAT που είναι ε, μια ομάδα που απαρτίζεται από διάφορους εταίρους, από συνδέσμους των κρατών μελών. Ε, είναι μια ομάδα εργασίας ε, για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και Φυσικά είναι διασυνοριακό εξορισμού το ηλεκτρονικό έγκλημα σε αντίθεση με άλλες μορφές εγκλήματος, άρα χρειάζεται διασυνοριακή ε, συνεργασία και όχι να περιμένουμε να οριμάσει η έρευνα, η ανάκριση σε ένα κράτος μέλος και μετά να ειδοποιήσουμε την ε, Europol. Εδώ μπορεί να υπάρξει κάποια σύγκρουση. Ε, η προληπτική εξουδετέρωση από τη μια και η συστηματική δίωξη και ανάκριση και έρευνα. Εδώ συγκρούνται οι απόψεις ε, και οι έννοιες. Χρειάζεται λοιπόν μια νομική σαφήνεια και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να ξεκολουθούμε με τα ευρήματα εδώ. Ποια είναι τα νομικά προβλήματα και δυσκολίες και οι προκλήσεις. Το ηλεκτρονικό έγκλημα πολλές φορές χρειάζεται ταχύτητα στην αντιμετώπιση του, αν θέλεις να συλλέξεις στοιχεία. Άρα τα πλαίσια που υπάρχουν για τη συνεργασία που είναι συμφωνίες για αμοιβαία δικαστική συνδρομή ε, είναι πάρα πολύ βαριές διαδικασίες, πάρα πολύ βραδίες και η τεχνολογία έρχεται να περιπλέξει τα πράγματα και πρέπει να επιταχύνονται και οι διαδικασίες. Ούτε εγώ, ούτε η οργάνωσή μας, ούτε ε, διεθνείς οργανισμοί θεωρούν ότι αυτό ευσταθεί. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία και περισσότερη πρόσβαση σε προφορίες που έχει ιδιωτικό τομέα. Πριν από λίγα χρόνια, στις πρώτες εκθέσεις του Κέντρου Αντιμετώπισης του ε, Εγκλήματος, είπαν ότι διστάζουν να το αναφέρουν οι διοκτικές αρχές, μεταξύ άλλων, και για λόγους γοήτρου ή φήμης. Θα πρέπει να ε, αναζητούν πολλές φορές τα στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι από ιδιώτες, από παρόχους εδώ υπάρχουν ζητήματα λοιπόν δικαιοδοσίας ε, και με τον εύλογο χρόνο που χρησιμοποιείται μέχρι να εκδικαστεί κάτι. Ας πούμε, αν ένα τέτοιο αίτημα κάνει τις εταιρείες να παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα, είναι πάρα πολύ προβληματικό. Άρα χρειάζεται να υπάρχει ένα ενημερωμένο νομικό πλαίσιο. Πριν ληφθούν οποιαδήποτε άλλα μέτρα πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Η νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και για την διαχείριση δεδομένων για προστασία. Υπάρχουν συμβάσεις και η σύμβαση της Βουδαπέστης η οποία δεν είναι προβληματική. Αυτό που έχει πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ε, καθορίσει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας και ζωής κάθε φορά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ευρήματα. Ποιες είναι οι συστάσεις τώρα της μελέτης. Τρεις ε, αναγράφονται εδώ και θα τις υπογραμμίσω. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αναθεωρηθούν οι δομές και εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ηλεκτρονικό έγκλημα, ε, συνεργασία με τις τρίτες χώρες, με, μάλλον με τρίτα μέρη, που μπορεί να είναι χώρες ή ιδιωτικοί φορείς, ε, θα πρέπει να γίνουν αναλογικά και να συνοδεύονται από όρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους όρους της αναλογικότητας, όπως ε, έχει να κάνει και τα ορίζει και η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας. Και τρίτον, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόφαση η δικαιολογία το ηλεκτρονικό έγκλημα ε, για να υπονομεύονται ε, πρωτόκολλα ασφαλείας ε, των πληροφοριών μεταξύ αυτών κρυπτογράφηση και ανωνυμοποίηση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε τη δόκτωρα ε, Βάντερ Μέρλεν και άλλα ομιλητή που θα μας παρουσιάσει την παρουσίαση για την ασφάλεια ε, στον κυβερνοχώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής διερεύνηση των κινδύνων και εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, and also... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε τη μελέτη μας Πολύ γρήγορα θα κοιτάξουμε τους βασικούς στόχους της μελέτης, τα βασικά πορίσματα και τις επιλογές πολιτικής που έχουμε αφορήσει. Ποιος είναι ο στόχος μας. Θέλουμε να εντοπίσουμε τις βασικές απειλές στον κυβερνοχώρο, τις βασικές δυνατότητες ε, αντιμετώπισης των προβλήματων ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις βασικές δυνατότητες της ΗΠΑ επίσης. Ταυτόχρονα θέλουμε να αποτιμήσουμε το πώς έχει η διασυνοριακή συνεργασία αυτή τη στιγμή και να δούμε και ποια είναι η αντίληψη για την αποτελεσματικότητα της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν να σας πω ποια είναι τα βασικά μας απορίσματα για τις απειλές, τις δυνατότητες, την συνεργική συνεργασία και την αντίληψη περί αποτελεσματικότητας. Ποιες είναι οι βασικές απειλές. Είναι ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από την πρώτη παρουσίαση σε αυτή την συνεδρίαση για τις ε, μελέτες ΑΙΟΚΤΑ της Europol. Εντοπίσαμε δύο πράγματα πρώτα απ' όλα εν μέρη, διότι θέλαμε, θέλαμε να είμαστε σαφείς. Η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την αποτίμηση των απειλών δεν είναι πάντοτε αυτή που θα θέλαμε. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται στην αποτίμηση των απειλών, αλλά δεν είναι η μόνη επιλογή. Οι Τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από μελέτες όπως η ΑΙΟΚΤΑ είναι κάποτε ασαφή. Δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ των πλαισίων αναφοράς. Τι είναι ε, απειλή, εργαλείο, όλα αυτά ε, υπολογίζονται από κοινού. Δεν υπάρχει σαφής ορισμός δηλαδή για το τι ακριβώς αναζητούμε. Κάποιες ε, μπορεί, για κάποιους το ίδιο πράγμα μπορεί να είναι εργαλείο, για κάποιους άλλους είναι απειλή. Ε, την ίδια οπτική γωνία την έχουμε συμπεριλάβει στην μελέτη. Δηλαδή ότι η αντίληψη για το τι ε, αποτελεί απειλή εξαρτάται από τα ποια εργαλεία χρησιμοποιεί ο καθένα. Και επίση τα αποδεκτικά στοιχεία μέχρι τώρα, τα δημοσιεύματα και οι σχετική βιβλιογραφία δείχνουν ότι διαφέρει η αντίληψη τη πολιτική. Αν μιλάμε για το τι προβάλλουν τα μέσα μαζική ενημέρωση ή τι αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί. Έτσι, ο στόχο ήταν να κάνουμε μια πρόταση για το πώ μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πιο εναρμονισμένο πλαίσιο για την αξιολόγηση, την αποτίμηση των απειλών. Για να είναι πιο σαφή και πιο αρμονική παντού. Ε, ο στόχος ήταν να μην υπάρχει επικάλυψη και ασάφεια για τις αρχικές πηγές που χρησιμοποιούνται. Εδώ λοιπόν αυτό είναι το πλαίσιο που θα θέλαμε να χρησιμοποιείτε και βλέπουμε ότι υπάρχουν πρώτα απ' όλα δράστες των απειλών, τα εργαλεία των απειλών που συνδυαζόμενα μπορεί να αποτελούν μαζί απειλή με σκοπό την καταστροφή, την ε, μη επιτρεπόμενη πρόσβαση και μετά υπάρχει και ο στόχος ε, και επίσης μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και άλλα στοιχεία όπως τον παράγοντα απειλή ή την συγκεκριμένη επίθεση. Αλλά ο στόχος είναι να εμπνεύσουμε την δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου. Συνεχίσαμε λοιπόν εδώ γιατί θέλαμε να πούμε κάτι επί της ουσίας για τις ε, κυβερνοαπειλές και συνεχίσαμε παρόλες τις δυσκολίες και τα παγρευτικά που αντιμετωπίσαμε. Βλέπετε ότι μεταξύ των παραγόντων της απειλής αναφέρονται πολύ συχνά οι ε, τα κράτη και οι κυβερνοεγκληματίες. Επίσης βλέπουμε να υπάρχει μια βιομηχανοποίηση του κυβερνοεγκλήματος, ε, μαζικοποίηση, δηλαδή η, αγορά, η μαζική αγορά υπηρεσιών και σε ό,τι αφορά τα εργαλεία των απειλών, συνήθως ε, το δόλιο ε, λογισμικό είναι από τα πιο χαρακτηριστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Αλλά είναι πολλά τα λογισμικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς τέτοιου είδους το λεγόμενο malware, το δόλιο λογισμικό, είναι ε, πολύ σχετικό πώς ε, λειτουργεί τελικά σε σχέση με το επίπεδο ασφάλειας και προστασίας από αυτό. Πώς μεταφέρονται λοιπόν όλα αυτά και πώς μεταφράζονται στις δυνατότητές μας να εξασφαλίσουμε κυβερνοασφάλεια. Έχουμε τρεις στρατηγικούς στόχους από την, Ευρωπα... από την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια. Έχουμε επικεντρωθεί στην αντικτικότητα, το κυβερνοέγκλημα και την κυβερνοάμυνα. Ε, βλέπουμε τι δυνατότητε υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ του οργανισμού και βλέπουμε ότι ω προ την αντοχή κατά του εγκλήματο έχουμε το, την ΕΝΙΣΑ, τον Οργανισμό για τα Δίκτυα και την Ασφάλεια των Πληροφοριών, που ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι δραστηριότητε κάποιων κεντρικών υπολογιστών και ε, εφόσον κάποια κάτι μέλη δεν έχουν σχετικό πλαίσιο, τα βοηθάει να το εγκαταστήσουν. Για το έγκλημα νομίζω με την Europol ε, καλύψαμε διεξοδικά το θέμα. Και στην κυβερνοάμυνα βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τόσο μεγάλε προσπάθειε, γιατί συνήθω πρόκειται για θέματα εθνική ασφάλεια, αλλά υπάρχει ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2014. Και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό τη Άμυνα στον κυβερνοχώρο στηρίζει την ε, ε, σωστή υλοποίηση αυτή τη στρατηγική. Μέρος της μελέτης ήταν και η σύγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ, που είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό τους, πολύ πιο περίπλοκο και με πολύ πιο μακρά ιστορία αντιμετώπισης του εγκλήματο. Η διαστρωμάτωση των οργανισμών και των φορέων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα είναι πολύ πιο ε, σύνθετη. Υπάρχει πολλή κουβέντα για την ε, ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ και παρά τις πολλές προτάσεις και αλλαγές που προβλέπονται, οι προσπάθειες ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί και εν μέρη διότι μπορεί να υπάρχει σύγκρουση με την αντίληψη περί θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη κυρίως. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα διάγραμμα, δεν είναι διεξοδικό, για τους φορείς των ΗΠΑ που ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια. Βλέπετε τα υψηλότερα επίπεδα, αλλά σας δίνω τουλάχιστον μια γενική εικόνα για το πόσες υπηρεσίες και φορείς εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Ως προς την ανθεκτικότητα λοιπόν, το Υπουργείο Εσωτερικών ασχολείται με αυτά τα θέματα, παίζει κεντρικό ρόλο. Γίνεται βέβαια πολλή κουβέντα για το ποιος θα πρέπει να έχει τον ηγετικό, τον κατεξοχήν ηγετικό ρόλο εδώ. Η οι επιμέρους υπηρεσίες ασφάλειας ε, που υπάγονται στο Υπουργείο πολλές φορές ακούγονται. Υπάρχει το Ομοσπονδιακό Γραφείο, το FBI, και οι μυστικές υπηρεσίες που υπάγονται στο ίδιο Υπουργείο ούτως ή άλλως. Ως προς το κυβερνό έγκλημα είναι κυρίως το Υπουργείο Άμυνας υπεύθυνο και η πολιτική στρατηγική φέτος εξέφραζε ρητός το πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητές τους περί Άμυνα. Ε, επόμενη διαφάνεια. Εάν περάσουμε από αυτές τις δύο γεωγραφικές ζώνες και δούμε την διακρατική συνεργασία, την διασυνοριακή συνεργασία, είναι σαφές ότι είναι καθοριστική σημασία σε αυτή. Και στις παρουσιάσεις που ακούσαμε προηγουμένως. Ε, έχει δοθεί έμφαση σε κάποιες μονομερείς ε, πρωτοβουλίες συγκεκριμένων εταιριών που δείχνουν όμως ότι αν δεν συνεργαστεί κανείς και ε, αν δεν υπάρξει συνεργασία πολιτικού και ιδιωτικού τομέα μπορεί τελικά να πληγεί η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Έχει νόημα λοιπόν η διακρατική συνεργασία προκειμένου να μην υπάρχουν συγκρόμενες δράσεις. Επίση, μόλι ακούστηκε ότι η αμοιβαία νομική αρρωγή και η σχετική διαδικασία έχει, ε, έχει θεωρηθεί παροχημένη και δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι αποτελεσματική. Αναφέραμε μία μελέτη που έγινε από το Κέντρο των Διεθνών Στρατηγικών Μελετών και εξευρέθηκε ότι Κάποιε υποθέσει, προκειμένου να ολοκληρωθούν στην έρευνά του, απέτησαν χρόνια αντί για μήνε. Αυτό ε, είναι ένα σε μάχη πώ θα τερμινεύσουμε. Βεβαίω η βασική πρόκληση, όπως προηγουμένως ακούστηκε, είναι να βρούμε μια λειτουργική ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων των ανακρίσεων και ερευνών και της διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα και είδαμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την τήρηση των δεδομένων. Η απαντήσεις που είχαμε μας είπαν ότι δεν μπορούσαν οι ερευνητές και ανακριτές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους εξαιτίας αυτού του νόμου. Επίσης χρειάζεται καλύτερη αναρμόνιση των πολιτικών μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη ροή πληροφοριών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και διεκτικών αρχών καθώς και εισαγγελιών. Πού μας οδηγεί λοιπόν αυτό προς την αποτελεσματικότητα. Οι δυσκολίες με την αποτελεσματικότητα, τα απαγορευτικά όρια είναι δύσκολο να καταματρηθούν λόγω της, σε, ε, της μεταβαλλόμενης απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα διαμορφώνεται. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρόσφατα κατέληξαν ε, σε συμφωνία για την ε, οδηγία νης και ήδη οι διαβουλεύσεις αυτές κράτησαν πάρα πολύ καιρό μέχρι να φτάσουμε εκεί. Υπάρχει ακόμη λοιπόν σοβαρό κατακαιρματισμό μεταξύ τη λειτουργία των διαφορετικών φορέων και συνολικά τη προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν τάσει βελτίωση. Η ελλείψεις ε, αποτελεσματικότητας στη διαφορετική ιεράρχηση των στόχων των κατων μελών είναι μια πρόκληση. Η οδηγία νης ναι, θα μας βοηθήσει να το ξεπεράσουμε, αλλά είναι ένα κρίσιμο σημείο αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις στην αποτελεσματικότητα. Ως την ομοθετική προσέγγιση υπάρχει μια αλλαγή από την εθελούσια συμμετοχή και την επίσημη στην δεσμευτική και ανεπίσημη. Αυτό έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στην πορεία μας για το μέλλον πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και σε ό,τι αφορά την σύγκριση με τις ΗΠΑ, αυτό που σημειώσαμε, συγκρίνοντα το τι συμβαίνει στην Αμερικανική πραγματικότητα, είναι ότι όλη η συζήτηση για την κυβερνοασφάλεια και τι νομοθετικέ προτάσει είναι πολύ περισσότερο προβεβλημένη στο κοινό. Υπ' αυτήν την έννοια θα πρέπει να, να παραδειγματιστούμε από τι ΗΠΑ. Διότι εκεί τα πράγματα αυτά συζητιούνται πολύ περισσότερο και σε επίπεδο μέσων μαζική ενημέρωση και ε, μπορεί να υπάρχει και καλύτερη ανταπόκριση από τον κόσμο. Επόμενη διαφάνεια οι πολιτικές επιλογές μας είναι ότι θα ενθαρρύναμε την ενίσα Μάλλον θα ενθαρρύναμε να υπάρχει καλύτερη εναρμόνιση των ε, αποτιμήσεων των απειλών με ένα κοινό πλαίσιο και με κοινού βασικού όρου. Έτσι θα είναι σαφέ το τι εννοούν οι μεν και οι δε και πώ οι διάφοροι φορεί μπορεί να ενισχύσουν ένα τον άλλο. Δεύτερο σημείο, θα ε, καλούσαμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο αμερικανικό παράδειγμα, ώστε να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσε υποδομέ όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό. Ε, Βεβαίω το EC3 ε, προβλέφθηκε για να καλύψει τα κενά, όμω υπάρχει τάση να προβλέπουμε νέε υποδομέ ενώ δεν χρησιμοποιούνται επαρκώ οι, οι, οι, οι τωρινέ. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό αυτό. Όπως είπα, ε, πετέχεται συμφωνία για την οδηγία νης, για την ασφάλεια των των πληροφοριών, αλλά μπορεί και να προκληθεί μεγαλύτερος κατακαιρματισμός. Επειδή δεν έχει προβλεφθεί η κατανομή, η ανταλλαγή πληροφοριών στην υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων. Από ό,τι ξέρω, προτάσει για την οδηγία, βάσει των πηγών μου τουλάχιστον, γιατί αυτά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν έχει προβλεφθεί αυτό που έλεγα. Δεν έχει περιληφθεί. Θα ήταν καλό να συμβεί για να προχωρήσουμε στη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κανονισμός της Europol βρισκόταν σε εξέλιξη όταν ε, εμείς εκπονούσαμε την ε, μελέτη μας και είχαμε κάποιες αποκρίσεις από τον ιδιωτικό τομέα για τα συμπεράσματά μας και όταν καταρτίζαμε το κεφάλαιο για τις πολιτικές επιλογές. Εγώ κοιτάξα πολύ σύντομα το κείμενο και είδα ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπου είναι δυνατόν να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά ε, ο κανονισμός ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. Τελευταία παρατήρηση έχουμε εντοπίσει συνειδητοποίηση, όπως ε, και περισσότερα θεσμικά όργανα, ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα ε, επιδόσεων μεταξύ των κρατών μελών, διαφορετικές δυνατότητες. Εάν θέλουμε όλα αυτά κάπως να ομογενοποιηθούν, πρέπει να τα εντοπίσουμε σωστά και να δούμε με τι εργαλεία, με τι μέσα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε για να καταμετρούμε σωστά έπειτα και την πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Έχουμε κάποια λεπτά για ερωτήσεις και για σχόλια θα απευθυνθούν προς το πάνελ. Ο κ. Μπόνι. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε επί θεμελιωδών ζητημάτων. Αν μιλάμε για έλλειψη εναρμόνισης, σε κάποιους άλλους τομείς προχωράμε όπως η οδηγία για την ασφάλεια των πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι ένα βήμα προς αυτή κατεύθυνση. Θα ήταν πολύ χρήσιμο εμείς σαν ευρωβουλευτές να έχουμε την άποψή σας για ποιους τομείς θεωρείται ανεπαρκής που υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αναφέρατε την ανάγκη μεγαλύτερης ε, ε, συνεργασίας Europol και και των άλλων μονάδων της ε, Ευρωπόλ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Είναι θέμα καλύτερης διαχείρισης, καλύτερης οργάνωσης ή θέμα πλαισίου. Τρίτον, Τι νομικές αλλαγές χρειαζόμαστε. Κάποιοι από εμά είπαμε ότι χρειαζόμαστε μια ασφάλεια δικαίου, νομική σαφήνεια. Θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες. Σε ποιους τομείς, πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Αναφέρθηκε επίσης ότι εξαιρετικές λύσεις για το θέμα της κρυπτογράφησης δεν είναι κάτι που απαιτείται. Χρειάζεται κρυπτογράφηση σε πολλούς τομείς από ό,τι καταλαβαίνω όσο υπάρχουν εξελίξεις στον ψηφιακό κόσμο. Απ' την άλλη πρέπει να βρούμε μια λύση ισορροπημένη. Έχετε κάποιες προτάσεις. Αν εμείς οι ευρωβουλευτές συζητούμε αυτούς τους τομείς βλέπουμε ότι πρέπει να δώσουμε κάποια μάχη και χρειάζεται να έχουμε τεχνογνωσία, άρα χρειαζόμαστε τη σοφία σας από αυτό. Μήπως μπορούσατε να μας πείτε τι σχέσεις πρέπει να έχουμε με τις τρίτες χώρες. Περιγράψατε τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΕΠΑ. αλλά έχουμε και τις χώρες της ανατολικής ε, γειτονίας. Πώς θα συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες. Τέλος. Επεσκέφθην την Ενίσα. Για τρία-τέσσερα χρόνια ο προϋπολογισμός παραμένει στη διαπίπεδα για την Ενίσα. Δεν ήθελα να αναφέρω και την Ευρωπόλ. Ίσως η ίδια κατάσταση να επικρατεί. Αν θέλουμε πραγματικά να καταπολεμήσουμε το ηλεκτρονικό έγκλημα, θα πρέπει να θεσπίσουμε ένα καλύτερο νομικό πλαίσιο. Πρέπει να καθορίσουμε τους στόχους μας και να δημιουργήσουμε το κατάλληλο δυναμικό, τις κατάλληλες δυνατότητες, να απασχολούμε τα κατάλληλα ε, άτομα και να υπάρχουν ε, τα χρήματα για να λειτουργούν σωστά αυτοί οι φορείς. Τέλος. Για τη μονάδα αυτή που αναφέρατε, που θα ξεκινήσει να λειτουργεί στην Ευρωπόλ, που σχετίζεται περισσότερο με θέματα τρομοκρατίας, που θα ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας από 1η Ιανουαρίου Μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Αν είστε έτοιμοι, τι χρειαζόσαστε. Υπάρχουν τρεις εβδομάδες ακόμα που πρέπει να διανύσουμε μέχρι να ξεκινήσει εργασίες η, μονάδα. Συμφωνώ με αυτό που είπατε κύριε Μπόνη για την Ενίσσα. Για... Έχω κάτι και εγώ να ρωτήσω για την κρυπτογράφηση. Όταν κάναμε τη συζήτηση για τη μαζική παρακολούθηση, συζητήσαμε και την κρυπτογράφηση. Μπορείτε να μας αναλύσετε το νομικό πλαίσιο γι' αυτό. Κάτι που έθιξε ο κ. Μπόνι. Ζητήσαμε από τους παρόχους πότε θα προβούν σε αυτή την κρυπτογράφηση για να παράσχουν την προστασία ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών. Οι αρχές τι άποψη έχουν γι' αυτό, τι πλαίσιο οικοδομείται γι' αυτό. Και ε, δεν θα είναι ποτέ τέλεια κρυπτογράφηση. Πού βρισκόμαστε, είναι πολύ αρχική η κατάσταση. Ρωτήσαμε και την Microsoft να μας πει τι δυνατότητες κρυπτογράφησης δημιουργούν πάνω σε αυτό. Η Άννα έχει το λόγο, λυπούμε. Ζητώ συγγνώμη. Δεν μπόρεσα να ακούσω τις αρχικές παρεμβάσεις Άκουσα όμως την κυρία Βαντερ Μέλεν και με επιβεβαιώνει στην αίσθηση που έχω ότι τα κράτη-μέρη μας κοροϊδεύουν ε, μας τους πολίτες, γιατί αν υπάρχει ένας κλάδος που χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση και από τον προϋπολογισμό ε, σε χρήματα αλλά και σε ανθρωπίνους πόρους, όχι μόνο οικονομικούς και στελέχωση, είναι κατεξοχήν αυτός πόσο σημαντικό είναι και κρίσιμο καταλαβαίνουμε για την ασφάλειά μας. Και δεν πιστεύω ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη θα υπάρξουν αυτές οι δυνατότητες, ούτε καν η βούληση για τις επενδύσεις και τις αλλαγές που χρειάζονται, εάν δεν υπάρξει μια υπερεθνική προσπάθεια για να γίνει κάτι τέτοιο. Και φυσικά δεν ε, δράσουμε από κοινού και με τρόπο συνεπή θα είμαστε τόσο ασθενείς όσο ο πιο αδύναμος κρίκος. Προχτές είχα ε, συμμετάσχει σε ένα δείπνο με εμπειρογνώμονες από διάφορα κράτη-μέλη και εταιρείε ε, που δραστηριοποιούνται στη ψηφιακή τεχνολογία και με όλα τα συμπαρομαρτούνται για την ασφάλεια και τα λοιπά στον κυβερνοχώρο και μου έλεγαν οι ίδιες εταιρείες και οι πόσο ήταν ε, μάρτυρες και τα θύματα των εσωτερικών ε, τσακωμών και καυγάδων μεταξύ των εθεσμών στην Ευρώπη, δηλαδή μεταξύ της ΕΝΗΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε προκειμένου. Δεν αφαιρθήκατε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνης, που είναι και ένας άλλος οργανισμός που αναπτύσσεται, που θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, και ε, να αναπτύσσεται και να έχει ένα πλαίσιο δράσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ιδιαίτερα για το ηλεκτρονικό έγκλημα ε, και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών. Αυτό πώς συνδέεται. Συμμετέχει ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Οργανισμός ο στρατός, τα επιτελεία θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο για την ε, φύλαξη των ε, κρίσιμων υποδομών. Και τέλος. Πρόσφατα πήγαμε στην Κίνα, αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας εδώ της ΛΥΜΠΕ και αναφερθήκατε σε αυτό ότι συχνά συνδέεται το ηλεκτρονικό έγκλημα με χώρες, ε, τις Ηνωμένε Πολιτείες. Πήγαμε όμως στη Huawei, δεν ξέρω αν ξέρουν πολλοί Ευρωπαίοι. Γουά σημαίνει Κίνα και Huawei σημαίνει ευημερία. Φαντάζεστε να λέγανε τη Google by American ή America Iberales. Αυτό σημαίνει η Huawei εταιρεία. Ευημερία της Κίνας. Και πολλές κυβερνήσεις μας δεν κάνουν συμβάσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με μια εταιρεία τέτοια, σύντη τη Huawei. Ή μάλλον υπογράφουν, ενώ είναι τεράστιο το σκοτάδι που επικρατεί εκεί. Και ξέρετε πώς είναι το κινέζικο σύστημα. Μήπως είμαστε εμείς οι ίδιοι ο χειρότερος εχθρός μας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε αυτές τις ηλίθιες πολιτικές λιτότητας που καταστρέφουν ε, ε δομές κρίσιμες για ε, την ασφάλειά μας, για να μην μιλήσω και για την ε, όχι αμυντική αλλά την επιθετική πλέον ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είσαι Σιλ Κέγγε, θέλεις, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω και σε σχέση με την αρμοδιότητα που θα αναλάβει η Europol μελλοντικά για την τρομοκρατία. Έχετε στα χέρια σας συγκεκριμένα νομικά μέσα για να καταπολεμηθεί για να καταπολεμηθούν οι περιπτώσεις εκφράσεις μίσους και τι σκοπεύετε να κάνετε στο πλαίσιο και στην περίπτωση της ριζοσπαστικοποίησης. Ευχαριστώ, Σεσίλ και γιατί πολύ γρήγορα θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ε, οι δύο εισηγητές μου έστειλαν ένα μήνυμα. Αλλά θα θέλαμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο γρήγορα. Θα πρέπει να πάρουμε το λόγο ευθύ αμέσω. Θα πρέπει πολύ γρήγορα να ακούσουμε του προσκεκλημένου ε, μα εδώ. Και επίση για το εργαλείο τη αμοιβαία ε, δικαστική συνδρομή. Το συζητάμε αυτό στο Κοινοβούλιο εδώ και ένα χρόνο και βρήκαμε ότι η Σύμβαση για το Εγκλήμα δεν αξιοποιείται επαρκώ. και ο μηχανισμός δικαστικής συνδρομή είναι πολύ αργός. Τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε αποτελεσματικότερα δικαστικά εργαλεία, αλλά λαμβάνοντας αφορμή και από όσα είπε ο κύριος Μπόνι. Ε, είναι πολύ σοβαρό θέμα και αγγίζει πάρα πολλά άλλα επιμέρους, με την ενίσα ας πούμε. Πρέπει να υπάρχει άμεση αντίδραση σε αυτές τις καταστάσεις. Και η Άννα Γκόμες συνήθως φέρνει και ένα καπεταπηγόντα χαρακτήρα στα ζητήματα που, σε που φύγουμε σε κάθε συζήτηση. Και παίρνω αφορμή και εγώ από αυτό. Βλέπουμε ότι οι πολίτες λόγου χάρη αισθάνονται ότι οι λογαριασμοί τους έχουν αποστραγγιστεί για να ε, αποφύγουμε μαζικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και ταυτόχρονα στρέφονται προς εμάς και μας ρωτάνε τι κάνουμε τελικά. Έρχεται εδώ η Europol και οι διάφοροι οργανισμοί να μας πούν τι κάναμε και θα πρέπει να σα ζητήσω συγγνώμη που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο για να ακούσουμε και τι απαντήσει σα. Ευχαριστώ όλους για τις παρουσιάσεις σα. Ήταν κάπως απρόσμενο το σημερινό απόγευμα. Σημειώστε αυτές τις ερωτήσεις. Εάν έχετε κάτι να πείτε, παρακαλώ να το πείτε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο όσον αφορά τις ερωτήσεις για το θέμα του νόμου. Πώς μπορούμε να πετύχουμε. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νόμους των κρατών μελών. Πρώτα απ' όλα για τη διατήρηση των στοιχείων. Υπάρχουν διαφορές Ακόμα και αποτελέσματα ερευνών δεν μπορούμε να τα στείλουμε σε κράτος μέλος, δεν μπορούμε να δώσουμε συνέχεια. Δεν ξέρουμε την άποψη της χώρας και κυρίως την, όσον αφορά την κακομεταχείριση των παιδιών υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, η νόμιμη ε, είσοδος στο λογισμικό, backdoors, οι, πάροχοι δίνουν ε, την κρυπτογράφηση στην ασφάλειά τους. Χρειάζεται όμως και μεθόδους παρακολουθήσεως των ε, στοιχείων ε, πριν κρυπτογραφηθούν. Οι ιδιωτικές αρχές χρειάζονται αυτό για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της κρυπτογράφησης. Αυτό πρέπει να γίνεται με δικαστική επιβλεψή. Το κάνουμε όμως για άλλα εγκλήματα γιατί όχι και για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Ανέφερα την υποχρεωτική αποκάλυψη στοιχείων Άλλες χώρες το προβλέπουν, άλλες όχι. Για τη συνεργασία των χωρών, με ποιες χώρες συνεργαζόμαστε, αναφέρω δύο, Ομοσπονδία της Ρωσίας και η Ουκρανία θα ήταν πολύ χρήσιμες, διότι κάποιες επιθέσεις που βλέπουμε και κάποιοι εγκληματίες προσπαθούν να κρυφτούν εκεί. Και η Europol δεν έχει δυνατότητα ανταλλαγή στοιχείων με αυτές τις χώρες. Για το θέμα της τελέχωσης που αναφέρατε, είχαμε διδοχικές κρίσεις Είχαμε κάποιες αυξήσεις του προπολογισμού για τους οργανισμούς και για την ε, Europol. Με τη μετανάστευση είδαμε ότι υπήρχε υποστήριξη αύξηση των πόρων, αλλά για το ηλεκτρονικό έγκλημα έχουμε 75 μέλη του προσωπικού, 17 προέρχονται από σημαντικό προϋπολογισμό. Η, τα άλλα στελέχη, άρα δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Για, τις, για τους λόγους και την τρομοκρατία δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε ξεκινήσει τα της τρομοκρατίας, δημιουργούμε αυτό το κέντρο που θα παρέχει υποστήριξη όσον αφορά τις έρευνες στο Παρίσι. Θα, θα έχουμε και τη μονάδα για το διαδίκτυο που θα συμμετέχει. Το ίδιο ισχύει, υπήρχε ισχυρή υποστήριξη από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο για να ανατεθεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά και ελπίζω το απόγευμα να συζητήσουμε και την ανάγκη για το περαιτέρω προσωπικό που απαιτούμε. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι μονάδες. Αυτά λοιπόν είναι είδη απαντήσω στις τεθήσεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Μην βιαζόσαστε, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο για να απαντήσετε. Ορίστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Νομίζω ένα από τα σημεία που πρέπει να διερευνήσουμε και που απασχόλησε και τους ε, βουλευτές είναι η σωστή εξισορρόπηση μεταξύ των αναγκών επιβολής του νόμου και των προστατευτικών που υπάρχουν για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αλλά αυτό είναι κάπως παραλογικό. Ισχύει μόνον εάν έχουμε ένα σαφές πλαίσιο που να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δίκαιων δικών της σωστής προσαγωγής, της σωστής προστασίας Αυτό είναι ένα θέμα και ποινικό και, και νομικό και πολιτικό. Προτού φτάσουμε σε τεχνικού χαρακτήρα συμφωνίες. Μετά το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τις περιοχές που εντοπίζει η μελέτη ότι χρειάζεται δράση για την ε, αμοιβαία νομική συνδρομή Υπάρχουν δυνατότητε βελτίωση. Έχουμε εντοπίσει αρκετέ περιοχέ όπου μπορούν να γίνουν βελτιώσει. Ένα άλλο βήμα, πολύ πιο φιλόδοξο, είναι να έχουμε την, το Ευρωπα... την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα ω βάση συνεργασία με διάφορε αρχέ και με τον ιδιωτικό τομέα αλλά και με άλλε χώρε. Στι Ηνωμένε Πολιτείε θα μπορούσαμε να έχουμε και εκεί έρευνε αν υπήρχε διατλαντική λόγω χάρη εντολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσει με έναν φιλοδοξότερο τρόπο. Ευχαριστούμε. Η δόκτωρ ε, Βαντεν Η κυρία Τζο, ίσως. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα απαντήσω μερικές από όσες τέθηκαν για τον κατακαιρματισμό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είδαμε από τη μελέτη μας ότι ακόμη και όταν υπάρχουν πρωτοβουλίες υψηλού επίπεδου που τις ε, οργανώνουν η ΕΝΗΣΑ και η ΣΥΤΡΙΑ, ε, λίγα ε, γίνονται επιχειρησιακά για τη συνεργασία εν τέλει. Σε ό,τι αφορά την κατανομή πληροφοριών και την οικοδόμηση δυνατοτήτων, έχουμε προσέξει ότι δεν υπάρχουν αρκετές συνομιλίες μεταξύ των όσων παίρνουν μέρος στις έρευνες στην πράξη και την ε, ε, ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο. Αυτό προέκυψε και από τις συνομιλίες μας με προσώπους των κρατών μελών. Ενώ γνώριζαν για την ΕΝΗΣΑ, έλεγαν ότι η συνεργασία τους με την ΕΝΗΣΑ είναι ε, η ελάχιστη δυνατή. Μάλιστα είναι και τελείως συγκυριακή. Αυτό δείχνει τι επίπεδο κατακαιρματισμού υπάρχει σε επιχειρησιακό επίπεδο. Έπειτα υπάρχει και διάτομα και ως ε, κατακαιρματισμός, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας που αναφέρεται και προηγουμένως, σωστά, λειτουργεί σε, ε, απομονωμένα, ενώ η κυβερνοασφάλεια και το κυβερνοέγκλημα συνήθως ε, χρήζουν κοινή αντιμετώπιση με τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Και θα έπρεπε να υπάρχει διατομιακή προσέγγιση. Στη μελέτη μας επίσης ασχοληθήκαμε και με τις συμφωνίες που έχουν προσωρινά εγκριθεί, αλλά οι διεκτικές αρχές λόγου χάρη δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται. Πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση των ε, ενδιαφερομένων και θα πρέπει κάτι να προβλεφθεί σχετικά στην οδηγία νης για να αποφύγουμε τον περαιτέρω κατακαιρματισμό και σε ό,τι αφορά τις ε, συνθήκες αμοιβαίας στήριξης, τα περισσότερα κράτη-μέλη προτιμούν τις διμερείς συμφωνίες ή τις πολυμερείς και αυτό μπορεί να έχει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά έχει και μειονεκτήματα. Ένα από τα σημεία που πρέπει να εντοπίσουμε είναι ότι, όπως είπε προηγουμένως και ο συνάδελφος, τα θέματα τα νομικά το τι νομοθετική πολιτική θα ακολουθήσουμε είναι σημαντικά. Αλλά για το κυβερνό έγκλημα ακριβώ πρέπει να ε, λάβουμε ειδική πρόβλεψη. Διότι η τεχνική διοργάνωση του κυβερνού εγκλήματος είναι πολύ διαφορετική από το του παραδοσιακού. Αυτές λοιπόν οι, λεπτομε... οι ειδικές ε, αυτά τα ειδικά στοιχεία του κυβερνού έγκληματο επιβάλλουν τέτοια αντιμετώπιση. Η συνάδελφο. Ε, ευχαριστώ για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και τις κρίσιμες υποδομές. Δεν ξέρω αν πρέπει να ασχοληθεί με αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Η κυβερνοανθεκτικότητα λόγω χάρη δεν είναι απαραίτητα διασυνδεόμενη με τις κρίσιμες υποδομές. Υπάρχουν βέβαια κρίσιμες υποδομές για την εθνική ασφάλεια, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα επιληθεί στο επίπεδο των κρατών μελών αυτό το θέμα. Αυτό είναι κάτι πάντως που καλό θα ήταν να συζητηθεί έπειτα ο συσχετισμό μεταξύ κρατών και εγκληματιών. Δύσκολο να απαντήσει κανείς αυτό, διότι απλώς υπάρχουν περισσότερο υποθέσεις και εικασίες εδώ. Δεν υπάρχουν αρκετά δημόσια νομικά έγγραφα. Η βιβλιογραφία δεν είναι αρκετά τεκμηριωμένη όπως θα θέλαμε. Ευχαριστώ πολύ και στους τέσσερις ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, συναρπαστική αυτή η συζήτηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους βουλευτές που παρέμειναν για τη συζήτηση αυτή, για την ανταλλαγή απόψεων. Δεν ξέρω να το πιστεύετε. Η Επιτροπή μας ε, πάντως έχει μεγάλες επιδόσεις ήδη για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Το έχουμε συζητήσει πολύ. Μην κοιτάτε σήμερα. Ε, θα επανέλθουμε, ε, όπως είπε και η κυρία Γκόμες, υπενήχθη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για τους πολίτες μας και θα επανέλθουμε. Και με διαρθρωμένο τρόπο γίνεται ο διάλογος και δεν είναι καθόλου αποσπασματικός και μεμονωμένος. Ευχαριστώ και πάλι. Πάμε μέσω στο σημείο 10 γρήγορα. Οι δύο συνεισηγήτριες ε, έχουν να κάνουν μια σύντομη ανακοίνωση. Δεν ξέρω ποια θέλει να ξεκινήσει πρώτη. Ρομπέρτα. Θες να αρχίσεις εσύ και μετά η Σεσίλ. Η Σεσίλ πρώτη. Πρόεδρε. Eh, ε, πρόεδρε, σημειώνω ότι θέλετε να συζητήσουμε το έγγραφο εργασία. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο την επόμενη Πέμπτη στο Στρασβούργο και είμαι βέβαιη ότι θα καλύψουμε τι διαφωνίε μα τότε υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες τις οποίες ε, συμφωνούμε. Μπορούμε να συμμεριστούμε και τα οκτώ έγγραφα εργασία και νομίζω ότι συμφωνούμε λίγο πολύ ε, και οι οκτώ σκεδεσηγητές. Λυπούμε απλώς που με αυτή την ευκαιρία είχα προσκαλέσει μια ομάδα φοιτητών από την Λουβέν, τους οποίους χαιρετώ και ευχαριστώ για την παρουσία τους. Απλώς να πω ότι είχαμε ανταλλαγή απόψεων πολύ χρήσιμη πριν την έναρξη της συνεδρίασής μας και αν συμφωνείτε πρόεδρε θα πρότεινα να τους ξανακαλέσουμε προκειμένου να παρευρεθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ όπου θα είναι ε, διαθέσιμα και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα και εκεί θα παρουσιαστούν. Υποθέτω ότι μιλάτε εκ μέρους και των δυο σα, ε, η Ρομπέρτα θέλει να πει κάτι. Λοιπόν, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε η Σεσίλ. Από την αρχή της ε, διαδικασίας έλεγα ότι πρέπει να πετύχουμε σύγκληση όλων των ε, πολιτικών ομάδων. Είχαμε την πρόθεση να παρουσιάσουμε δύο έγγραφα σήμερα, ένα για τη διαχείριση των συνόρων και ένα για την αποτελεσματική εφαρμογή του CEAS συμφωνίας. Δεν καταλήξαμε σε κάποια συμφωνία και του ΚΕΣΑ. Λοιπόν, και θα θέλαμε να μας επιτρέψετε σε άλλη περίσταση να έρθουμε να το συζητήσουμε, να παρουσιάσουμε τα έγγραφα, όταν θα έχουμε πετύχει συμφωνία, όταν θα έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό σύγκλησης, όλες οι πολιτικές ομάδες θα έχουμε συγκλίνει και πραγματικά ελπίζω ότι όλα αυτά θα είναι δυνατό να γίνουν πριν το τέλος του έτους στην συνεδρίαση που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ για τις εξηγήσει για όλα αυτά. Προφανώς θα επαναπρογραμματίσουμε την συνεδρίαση. Εξηγήθηκαν οι λόγοι. Ως Πρόεδρος, τώρα μόλις το έμαθα, ζητώ συγγνώμη από τα μέλη που ήρθαν συγκεκριμένα για το σημείο αυτό. Ελπίζω να μείνετε για το επόμενο σημείο στο οποίο θα αναφερθώ σύντομα. Ζητώ συγγνώμη σε εκείνους από εσά που, είδατε, που ήρθατε εδώ συγκεκριμένα αυτό το σημείο. Ελπίζω να κατανοήσατε την εξήγηση που έδωσαν οι συγγήτριες και τώρα είμαστε έτοιμοι για το σημείο 11. Θα διατρέξουμε την υπόλοιπη μερίσια διάταξη. Όλοι είναι κουρασμένοι, είναι πέμπτη απόγευμα, το καταλαβαίνω, αλλά έχουμε και άλλα σημαντικά σημεία και ερχόμαστε στο σημείο 11, μελέτη, σχετικά με τις συνεργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης που ανατέθη από το, τη Διεύθυνση Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το θεματικό τμήμα, και παρουσίαση γίνεται το καθηγητή. Α, αλλάξαμε. Α, γι' αυτό έκανες αυτά που έκανες. Για πες μου λοιπόν. Oh, somebody substituted. Uh, That's what was going. <laughs> My apologies. So yeah, um, Λοιπόν, η παρουσίαση, ο καθηγητής Φίλιπ Ντεμπρόικερ δεν είναι εδώ, διότι καθυστέρησε η πτήση του. Άρα, η δόκτωρ ε, Γκαρσία Αντράδε θα κάνει την παρουσίαση μόνη της. Εξηγήστε μας περί τίνος πρόκειται για τη μελέτη αυτή που αναθέσαμε, για την ολιστική προσέγγιση στη μετανάστευση. Θα μας τα εξηγήσετε όλα εσείς και μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις από τους συνεισηγητές και από τα μέλη. Παρακαλώ ξεκινήστε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πρόσκλησή σας. Είναι τιμή για μένα που παίρνω το λόγο εδώ. Ομιλούσα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών εκ μέρους της ομάδας ε, των ερευνητών που ανέλαβε τη μελέτη για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες στον τομέα της μετανάστευσης θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μας απαρτιζόταν από την υποφανωμένη τον Ιβάν Μαρτίν από το Ευρωπαϊκό ε, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, με τη συνδρομή του Βιώρικα Καβίτα και του Σέζιο Μανανασβίλη και την εποπτεία του καθηγητού Φιλίπ Ντεμπρικέρ από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και, ε, και, και την καθηγήτρια Χριστίνα Χορτάσαρ από Ουνιβερσιτάτ Ποντιφίσια Κομίλιας. Και ε, μέλος της Ισπανίας στο δίκτυο Οδυσσέους. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια, ο σκοπός και το πλαίσιο, το πεδίο εφαρμογή της μελέτης, το πλαίσιο που εξέτασε, καθορίστηκε από μια ανάλυση της γενικής στρατηγικής της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες στον τομέα της μεταναστεύσεως και του ασυλού, κάτι που ζητήθηκε από το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου της 17 Δεκεμβρίου του 2014, η προσέγγιση, η συγκεκριμένη προσέγγιση που ακολουθήσαμε εστιάστηκε επί της ε, υλοποίησης και αξιολογήσεως του πολιτικού πλαισίου που κατήφθηνε τη συνεργασία με τέτοιες χώρες στον τομέα αυτό και η σφαιρική προσέγγιση στην μετανάστευση στην κινητικότητα, η ΓΑΜ. Ε, λοιπόν, λήφθη υπόψη τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση η προσέγγιση αυτή. Πρέπει να εστιαστούμε τώρα σε μια ισορροπημένη, συνεκτική και αποτελεσματική υλοποίηση και εξολόγηση αυτών που έχουν επιτευχθεί. Τώρα, ποια είναι η σημασία της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Αυξήθηκε η σημασία της συνεργασίας πρόσφατα λόγω των προσφάτων γεγονότων που συνδέονται με τη μεταναστευτική κρίση και πιο συγκεκριμένα την προσφυγική κρίση και εν ώψη των προσφάτων εξελίξεων και θέτοντας στο πλαίσιο αυτό τη μελέτη, θα ήθελα να τονίσω τρεις ανησυχητικές τάσεις. Η πρώτη είναι ότι η επανεισδοχή και η διαχείριση των συνόρων φαίνεται να αναφέρονται εκ νέου στις συζητήσεις στην Ευρώπη, κυρίως υπό το φως ε, της συνεδριάσεως για τη διαδρομή της, των Δυτικών Βαλκανίων του Οκτωβρίου και του σχεδίου δράσεως ε, που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρειάστηκε αλληλεγγύη με τρίτε χώρε για να αντιμετωπιστεί η κρίση των προσφύγων σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση και φαίνεται ότι έγινε πιο καλά αντιληπτό ε, από πλευράς οικονομικής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχνώντα άλλα στοιχεία όπως είναι η μετεγκατάσταση και άλλη ενισχυτική τάση που είναι η αύξηση των ανησυχιών για την ασφάλεια στον τομέα μετά τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι. Τώρα, να σας παρουσιάσω εν συντομία την δομή και το περιεχόμενο της μελέτης. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εξωτερική διάσταση του ασύλου και της μετανάστευσης και επισκοπώντας εντάχει του θέματος της κατανομής μεταξύ των μελών των διαφόρων ομοδιοτήτων στον τομέα, το πρώτο τμήμα εξετάζει και αναλύει τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεργάσει σε τρίτες χώρες σε θέματα μεταναστεύσεως και ασύλου. Τα μέσα υποδιαιρούνται σύμφωνα με την φύση τους σε πολιτικά, εργαλεία όπως διάλογος διμερής και περιφερειακός για αυτά τα θέματα, συμπράξεις για κινητικότητα, κοινά θεματολόγια για αυτά νομικά μέσα όπως συγκεκριμένε συμφωνίες για τη μετανάστευση, επανεισδοχή, διευκόλυνση θεωρήσεων καθώς και ε, ρήτρε για τη μετανάστευση σε συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας και μετά διάφορα επιχειρησιακά εργαλεία δηλαδή προγράμματα περιφερειακής προστασίας, νέες εκδοχές, περιφερειακή ανάπτυξη και προστασία, διευθετήσεις Frontex και εξωτερικές δράσεις σε άσο. Αυτή η ανάλυση συμπεριλαμβάνει χαρτογράφηση των οικονομικών μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι διαφορετικά και απαραίτητα εργαλεία χρηματοδοτήσεως για τη συνεργασία με τέτοιες χώρες από την DG DEFCO, και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τις σχετικούς πόρους και μια σύντομη επισκόπηση των διαφόρων λεπτομεριών των διμερών συμφωνιών εξωτερικής συνεργασία των κρατών μελών. Στο δεύτερο τμήμα αξιολογούμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της χρήσης των εργαλείων αυτών, της εξωτερικής συνεργασίας για το άσυλο και τη μετανάστευση, από τριπτή προσέγγιση, αντίκτυπο όσον αφορά τους στόχους που επιδιώκονται, ουσιαστική διάσταση, Δεύτερον, ποιε είναι οι συνέπειε τη φύσεω των χρησιμοποιούμενων μέσων για του σκοπού αυτού, λειτουργική διάσταση δηλαδή. Και τέλο, οι διάφορε προκλήσει όσον αφορά το συντονισμό για την έγκριση και εφαρμογή αυτών, που αυτή είναι η θεσμική διάσταση. Και τέλο, παρουσιάζουμε συγκεκριμένε μελέτε για τη Μολδαβία, το Μαρόκο και την Τινησία, προσπαθώντα να δώσουμε μια εμπειρική εικόνα του θέματο που εξετάζουμε. Στο τρίτο τμήμα εκφράζουμε συμπεράσματα και προτείνουμε και συγκεκριμένες συστάσεις για μελλοντικές δράσεις και αυτό είναι το θέμα επί του οποίου θα επικεντρωθώ τα επόμενα λεπτά και λόγω χρονικών περιορισμών θα αναφέρω μόνο μερικές λεπτομέρειες. Ε, οι συστάσεις μας σχετίζονται με τα διάφορα πορίσματά μας. Πρώτα απ' όλα υπάρχει σαφής ανάγκη βελτιώσεως της οροπίας μεταξύ των διαφόρων συνιστοσών της σφαιρικής προσεγγίσεως για την κινητικότητα και τη μετανάστευση. Η ανάλυση των εργαλείων GAM και η εφαρμογή αυτών επιβεβαιώνει μια ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ των τεσσάρων συνιστοσών του GAM υπέρ του πυλώνα που αφορά την καταπολέμηση της παράτυπης μεταναστεύσεως που είναι ο πιο ολοκληρωμένος πυλώνας που εστιάζεται σαφώς στην επανεισδοχή και διαχείριση των συνόρων. Άρα υπάρχει μια ανάγκη να ενισχύσουμε την εξωτερική δράση της ΕΕ για την νόμιμη μετανάστευση ενισχύοντας το στόχο εντός των συμπράξεων για την κινητικότητα και χρησιμοποιώντας συμφωνίες σύνδεσης για αυτό το σκοπό, διότι τώρα αναγνωρίζουν μόνα δικαιώματα για τους νόμιμους μετανάστες που ήδη διαμένουν νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν αυτού, πέρα της μεγιστοποίησης της αναπτυξιακής διάστασης της μετανάστευσης, που είναι ένας πυλώνας που χρήζει προσοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τον πυλώνα για το άσυλο και τη διεθνή προστασία για την ώρα, ε, οι συμφωνίες ε, δημιουργούν δυναμικό με πολύ μικρή συνιστόσα της μετεγκατάστασης εξωτερική διάσταση της ΕΑΣΟ είναι υποανάπτυκτη λόγω περιορισμών δημοσιονομικών και λήψης πολιτικής βουλήσεως. Αυτή η ανισορροπία επίσης είναι αντιληπτή στην εφαρμογή των διαφόρων οικονομικών μέσων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτεί πρωτοβουλίε και προγράμματα συνεργασία με τίτε χώρε, παρόλο που υπάρχει σαφή συνεχή αύξηση των συνολικών δαπανών όσον αφορά τη δράση τη μετανάστευση τα τελευταία χρόνια, η χρήση των πόρων, πιο συγκεκριμένα να εστιαστούμε επί των πόρων ΔΕΦΚΟ, του, του, προγράμματος, του πρώην προγράμματος ενίας ή του προγράμματος μετανάστευσης του άσυλο επικρατεί η του προγραμματος μεταναστευσης του ασυλο επικρατει κατά καταπολεμηση της παράτυπης μετανάστευση και η νόμιμη μετανάστευση ε, και η ανάπτυξη δεν, παίρνουν, δεν, δεν έχουν τόσο μεγάλη προτεραιότητα. Όσον αφορά την συνοχή πολιτικής έχουμε ένα θετικό βήμα κατά την άποψή μας. Δηλαδή έχουμε συμπεριλάβει στο άσυλο μετανάστευση και το Ταμείο για την ένταξη των ιδιωτικής ε, θέμης εξωτερικές δράσεις συνεργασίας που πετυχαίνουν στόχο μετανάστευσης προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αντί πτυξιακή πόροι να πηγαίνουν προς αυτό το σκοπό όπως γινόταν πριν με τα άλλα προγράμματα. Τα εργαλεία ΓΑΜ της συνεργασίας και τα οικονομικά μέσα αυτά εστιαζόταν σε γεωγραφικά στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη και τον Νότιο Κάφκασο, τις χώρες των περιοχών αυτών. Μόλις πρόσφατα η συνεργασία έχει εντατικοποιηθεί με χώρες της Νοτία Μεσοχείου, τύπος Σαχάριας Αφρικής και χώρες Ανατολικής Αφρικής. Άρα χρειάζεται επανεξισορρόπηση γεωγραφική των γάμ. Δεύτερον, είναι απαραίτητο, θα έλεγαμε, να ενισχύσουμε την προσέγγιση της εταιρική σχέσης. Θα πρέπει όλο και περισσότερο να εμπλέκονται στην προσπάθεια και στη διαπραγματεύση του σχεδιασμού των μέσων ΓΑΜ τρίτε χώρε. Κάτι θα διευρύνει την φύση σύμπραξη των μέσων αυτών. Αυτό αφορά συμπράξει για την κινητικότητα και υπάρχουν ομοιότητες για τη δομή και ε, όσον αφορά τι συμπράξεις και δείχνει ότι δεν υπάρχει ε, σωστή διαπραγμάτευση με χώρες και το ίδιο με άλλες προσεγγίσεις όπου υπάρχει ε, έλλειψη ε, υιοθεσία από τους ντόπιου φορείς. Λοιπόν, χρειάζεται να τονώσουμε και την κινητικότητα, θα πρέπει να διευκολύνουμε ε, τις θεωρήσεις διαβατηρίων και θα πρέπει η κινητικότητα να είναι αυτόνομος σκοπός όταν η χώρα δεν θέτει κινδύνου, δημιουργεί κινδύνου όσον αφορά τον, την παράτυπη μετανάστευση και θα πρέπει να ξεκινήσουμε προβληματισμό σχετικά με το τι μπορούμε να προβλέψουμε στου εταίρου μα μετά την επιτυχή λήξη ενό διαλόγου για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για να διατηρηθεί η όλη ορμή και η βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί. Η πολιτική επανεισδοχή από την πλευρά τη θα πρέπει να εστιάζεται επί των χωρών προελεύσεω για να αποφύγουμε δυσκολίε μακροσκελεί διαπραγματεύσει και αναθεωρήσεις ε, όσον αφορά τις χώρες διέλευσης και η ρήτρα τρίτης χώρας της Συμφωνής Επανεισδοχής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο με σημαντικές χώρες διέλευσης υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο ενισχύσεων και βοηθείας. Τρίτον, σημαντικότατο ζήτημα. Α, συγγνώμη, δεν είπα ότι θέλω την επόμενη διαφάνεια. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Λοιπόν, όσον αφορά εξορθολογισμό και την αύξηση του συντονισμού. Λοιπόν, καταρχά να πω ότι ο πολλαπλασιασμό των περιφερειακών διαλόγων περί μεταναστεύσεων, πολλές χώρες συμμετέχουν ταυτοχρόνω σε αυτού, απαιτεί βεβαίως βεβαίως εξορθολογισμό και περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις πρακτικές και επιχειρησιακές αξίες και τιμές της συνεργασίας αυτής. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα χρηματοδοτήσεων από διάφορε πολιτικέ, από εσωτερικών, αναπτυξιακή συνεργασία, πολιτική γειτονία, που ανταποκρίνονται σε συγκρου... αντικρουόμενε λογικέ που ακολουθούνται και καμιά φορά αυτό οδηγεί σε επικαλύψει και αυτό παρεμποδίζει βεβαίω την ορατότητα, τη συνοχή και το δημοκρατικό έλεγχο των όσων πράττονται. Άρα θα ήταν ευκταίο να απλουστευτεί το όλο οικονομικό πλαίσιο από πλευρά λειτουργική διάφορα πολιτικά εργαλεία είναι και πιο κοινά, που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην εξωτερική διάσταση και θα ήταν ίσως χρήσιμο να ξεκινήσει η συνεργασία, όμως εν ώψη των κενών του υπείου δικαίου soft law θεωρούμε ότι αυξανόμενη ε, προσφυγή σε πιο, σε πιο αυστηρό δίκαιο χρειάζεται για να δίνονται, να τηρούνται οι δεσμεύσει, να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των μεταναστών σε τομεί όπω είναι η εισδοχή, η ένταξη και η κοινωνική ασφάλιση. Οι προκλήσει είναι μεγαλύτερε, θα έλεγα, σε θεσμικό επίπεδο. Ε, Καταρχά, όσον αφορά τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το συντονισμό αυτών, θα έλεγα τα κράτη-μέλη μεν επιμένουν να εμπλέκονται σε κάθε δράση Έχουμε δει όμως με τη μελέτη μας ότι δεν εξασφαλίζουν πάντα τη συμμετοχή τους εκ των υστέρων στα διάφορα εργαλεία ΓΚΑΜ, όπως είναι ο περιφερειακός διάλογος ή τη συνέχεια που δίδεται στις συμπράξεις κινητικότητας. Επίσης υπάρχει έλλειψη συστηματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 100 μελών σχετικά με τα όσα γίνονται σε διμερές επίπεδο και λόγω της υποχρεωτικής φύσεως της αρχής θεμητής συνεργασίας θα ήταν καλό να έχουμε κάποια προδιαγραφή δευτεροβάθμι, δευτεροβάθμιας νομοθεσίας για να τα εξασφαλίζουμε αυτά και να συμπεριλαμβάνονται ρητέ ε, υποχρεώσεις για ανταλλαγές πληροφοριών, διμερεί συμφωνίες και προγράμματα, να συζητούνται τα σχετικά μέτρα και να εξασφαλίζεται ο εσωτερικό συντονισμό πριν να υιοθετηθούν αυτά τα μέτρα. Και σχετικά με αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η προστιθέμενη αξία των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε σχέση με τις διμερείς δράσεις των κρατών μελών, ποια είναι. Θα ήταν καλό να να καταργηθούν οι ρήτρε συμβατότητα τη Συμφωνία Επανεισδοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπουν την εφαρμογή επιστροφών μέσω υφισταμένων επισήμων ή ανεπισήμων διευθετήσεων των κρατών μελών. Αν αυτή η ρήτρα καταργηθεί, αυτέ οι ρήτρε καταργηθούν, θα εξασφαλίσει τη μειούμορφη εφαρμογή των συμφωνιών τη Ευρωπαϊκή Ενώση περί επανεισδοχή. Έτσι, θα εξασφαλίζεται η προστιθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ενώσης όσον αφορά τι ε, αυτέ τι συμπράξει και θα δίδεται η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής σε πολυμερείς συμφωνίες και προγράμματα που εκεί που εμπλέκονται πολλά σε συνεργασίες ε, ε, κινητικότητας και όχι μεμονωμένα Όσον αφορά τη θεσμική διάσταση, και τον διοργανικό συντονισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλω την προηγούμενη διαφάνεια παρακαλώ. Όσον αφορά το διοργανικό συντονισμό, αρκετοί εμπλεκόμενοι, οι περισσότεροι από αυτούς συμφωνούν ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που συμμετέχει στην εξωτερική διάσταση θα πρέπει να αυξηθεί, αλλά για να επιτευχθεί αυτό για αυτό το σκοπό ε, η, η, δυναμι, η δυναμικότητά της να αυξηθούν και η χρηματοδότηση και χρειάζονται και αξιωματικοί σύνδεσμοι στις αντιπροσωπήσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να δρουν σαν βασική πολιτική υποστήριξη παρέχεται επιτόπου για την εφαρμογή των ΓΑΜ Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου στην εξωτερική διάσταση της μεταναστεύσεως και του ασύλου όπως θα δούμε στο θέμα του ελέγχου και της αξιολόγησης ε, μετά. Όσον αφορά το διοργανικό συντονισμό στο επίπεδο αυτό θα έλεγα ότι πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη αυξήσεως του συντονισμού όσον αφορά τις συγκλίνουσες προτεραιότητες μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπλέκονται στην εξωτερική διάσταση DEFCO, NEAR και HOME, οπότε θα είναι σημαντικό καθήκον αυτό για την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντός του Συμβουλίου θα ήταν καλό να δημιουργηθεί μια μονάδα επιφορτισμένη με το συντονισμό όλων των ομάδων εργασίας ε, και εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με την εξωτερική διάσταση ή να διευρυθεί ο συντονιστικός ρόλος της ομάδας υψηλού επίπεδου για το άσυλο και την μετανάστευση. Τελικά λοιπόν ε, το τέταρτο βασικό συμπέρασμα που βρίσκεται στην επόμενη διαφάνεια αναφέρεται σε μεγαλύτερη διαφάνεια για καλύτερη αξιολόγηση και έλεγχο ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε συντάσσοντας την μελέτη ήταν και το εξής προβλήματα που αφορούσαν την διαθεσιμότητα των πληροφοριών και την έλλειψη των προσπαθειών αξιολογήσεως κάτι που παρεμποδίζει συστηματική αξιολόγηση του αντιχτύπου και της αποδοτικότητας του ΓΑΜ. Επίσης την κατανομή των πόρων, την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων. Θα ήταν λοιπόν αναγκαίο περιοδικά να γίνεται μια πλήρης αξιολόγηση κάθε μέσου ΓΑΜ στα μέσα συνεργασίας και οικονομικά μέσα. Παράδειγμα, η προηγούμενη αξιολόγηση η εξολογήσει ε, για την επανεισδοχή ε, χρονολογούνται το 2011 και στην περίπτωση των συμφωνιών θεωρήσεις και συμφωνιών κινητικότητας χρονολογούνται εκθέσεις από το 2009. Όσον αφορά την αξιολόγηση των εφαρμοσμένων προγραμμάτων θα ήταν ευκταίο όχι μόνο να εστιαστούμε στα αποτελέσματα των προγραμμάτων και τον τακτικό χαρακτήρα των δαπανών και τη σωστή χρήση των δαπανών, αλλά και τι συνέπειε είχε το πρόγραμμα σε σχέση με του στατηγικούς στόχου του προγράμματο και σε σχέση με το γάμ και θεωρούμε αναγκαίο επίση τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να παρέχουν πλήρη ακριβή στοιχεία όσον αφορά την χρήση των μέσων γάμ που επιτρέπουν την πλήρη λεπτομερή αξιολόγηση αυτών, παραδείγματο χάρη ε, για τις επιστροφές θα ήταν απαραίτητο να τροποποιηθεί ο κανονισμός 862 του 2011 όσον αφορά στατικά στοιχεία περί μεταναστεύσεως και διεθνούς προστασίας, ούτως ώστε να απαιτείται από τα κράτη-μέλη να παρέχονται στατιστικά στοιχεία στο Eurostat όσον αφορά τις επιστροφές και αριθμούς ανθρώπων που επιστρέφονται και ομαδοποίηση κατά τα ομάδα ε, πράξης είναι συμφωνία επανεισδοχής, εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο ή διμερής ρύθμιση για εκείνους που επιστρέφουν, έτσι ομαδοποιούνται οι επιστρέφοντες, να ξέρουμε ποιο μέσο χρησιμοποιείτε και να μπορείτε να καθορίζετε και η χώρα επιστροφής, διότι τα στοιχεία δείχνουν μόνο την εθνικότητα εκείνου που επιστρέφει. Η αξιολόγηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει βεβαίως αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα των μέσων του ΓΚΑΜ, αν θεωρούμε παραδείγματο χάρη για ε, τις εξωτερικές δράσεις της Frontex για άλλα μέσα πώς χρησιμοποιούνται και τέλος στη μελέτη μας θεωρήσαμε ότι υπάρχει ανάγκη να βρεθούν τρόποι αυξήσεως του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία, όσον αφορά την εξωτερική διάσταση της πολιτικής, τη μετανάστευση και το άσυλο σχετικά όσον αφορά πολιτικά και περισσιακά μέσα τα οποία όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται στην εξωτερική διάσταση, τακτικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις όσον αφορά την έγκριση και ε, συμπράξεις ε, κινητικότητα, DPP, GAMS, εξωτερικές δραστηριότητες, Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οργανισμών αυτής, όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται συστηματικά σαν αναλύσεις εντός του Ευρωκοινοβουλίου και πέραν αυτού και συμπληρωματικά θα πρέπει ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διεθνείς συμφωνίες όπως συμφωνίες επανεισδοχής ε, συμφωνίες διευκολύνσεως θεωρήσεων δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην επίσημη ε, στο άρθρο 218 της συνθήκης για τη σύμφωνη γνώμη, όχι σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε να υθετηθούν μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής αυτών των συμφωνιών και πιο συγκεκριμένα τι αντίκτυπο έχουν στους μετανάστες. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Θα χαρά να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σύντομες ερωτήσεις, σχόλια. Η Σεσίλ Κέγκε, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την άριστη παρουσίαση. Συμφωνώ για πολλά από αυτά που μας αναφέρατε για την έρευνα. Έχω, είχα μια σειρά από ερωτήσεις, αλλά τελικά η ομιλήτρια ήταν τόσο καλή που αναπτύσσοντας την παρουσίασή της απήντησε σε όλα. Είναι σωστό να εκτιμηθούν διαφορετικά οι διαφορετικοί παράγοντε γιατί πρέπει να επικεντρωθούμε στην καταπολέμηση τη λαθρομετανάστευση. Αυτό πρέπει να προγραμμιστεί. Η ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων και πώ θα συμμετέχουν περισσότερο οι τρίτε χώρες γίνεται ζωτική σημασία. σω είναι κάτι που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο. Το τι γίνεται με τα αντίτιμα προ τα τρίτα κράτη το οποίο το σχολιάσατε καθώς μιλούσατε. Και τελευταίο σημείο που βρίσκω σημαντικό είναι οι πολιτικές επαναπατρισμού. Πώς συνεργαζόμαστε με τις χώρες προέλευσης για τις επιστροφές και αν μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές και ως προς αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ λοιπόν, αλλά σε γενικέ γραμμές συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που, συμπερι... που συμπεριλαμβάνει έτσι και το έγγραφο. Ευχαριστώ πολύ. Άλλα σχόλια. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη, παρακαλώ. μικρόφωνο, κυρία Σφινέλη, δεν δουλεύει το μικρόφωνο. Ε, δεν λειτουργεί το μικρόφωνο μου. Ε, Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ήθελα να πω ότι και εγώ θεώρησα ότι πολλά σημεία ήταν πέραν του ότι ήταν ενδιαφέροντα σημεία, με έβρισκαν και σύμφωνοι. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση επί της ουσίας ε, όσον αφορά το ρόλο που τα εθνικά κράτη και οι πολιτικές τους μπορούν να παίξουν σε αυτό το πλαίσιο. Το θέτω αυτό σαν ερώτημα διότι βλέπω ότι στην έκθεση βλέπουμε μεγάλο ρόλο για τη Frontex. Ένα ρόλο κατά την άποψή μου ε, πολύ λίγο, πολύ ανίσχυρο της ΕΑΖΟ και μετά μιλάμε για δράσεις εξωτερικές, κοινέ ευρωπαϊκές εξωτερικής δράσης. Όμως η εξωτερική δράση Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ε, κάτι το οποίο είναι καθοδόν, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί στην πολιτική, εξωτερική πολιτική ευρωπαϊκή, δεν έχουμε ακόμα δυστυχώς. Όσον αφορά λοιπόν την Frontex και τη δραστηριότητά της στο ΓΑΜ, θα ήθελα να επενθυμίσω την προσοχή πρέπει να δώσουμε σε κάτι. Υπάρχουν συμφωνίες, όπως η πρόσφατη που έγινε, που συνήφθη. Μεταξύ των 28 με την Ελλάδα, τη συμφωνία της 27ης Νοεμβρίου, όπου η παρουσία της Frontex στα σύνορα και ενδεχόμενη συνεργασία με τρίτες χώρες ήταν αποφάσεις που έπρεπε να ταιριάξουν με τις αποφάσεις των κρατών μελών. Υπήρχε κάποια αυτονομία των κρατών μελών. Τώρα όμως έχουμε επιστολή της Frontex που απεστάλλει σε όλα τα 28 κράτη-μέλη της Ενώσεως σε όλους τους υπουργούς της Ενώσεως και στην επιστολή αυτές οι συμφωνίες υποδιαιρέσεως των αρμοδιοτήτων δεν γίνονται σεβαστές. Δηλαδή οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν ένα της Ελλάδος όταν η Ελλάδα δέχτηκε να έχει την Frontex στα σύνορα δεν έγιναν, δεν εφαρμόστηκαν. Η ελληνική κυβέρνηση απάντησε λέγοντας αυτή τη θέση ότι αυτές ε, οι συνθήκες της συμφωνίας δεν μπορούν να, να ισχύσουν για τη Frontex σε κρίσιμα σύνορα της Ένωσης και την άποψή μου δεν μπορούν να λειτουργήσουν διότι αυτά τα αιτήματα της Ελλάδας που έγιναν δεκτά και απερίφθησαν μετά ήταν απόλυτα θέμητα σαν διεκδικήσεις και σαν απαιτήσει. Θα ήθελα την άποψή σας από αυτόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπάρπαρα. Θέλετε να απαντήσετε, δόκτωρ Αντράντε. Ναι. Επειδή άλλαζα γλώσσα, ε, δεν ε, κατάλαβα πάρα πολύ καλά την τελευταία ερώτηση. Επειδή ε, αλλάζω γλώσσες, αλλά ακούω από τα ακουστικά, δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά την τελευταία σας ερώτηση. Μπορείτε να την επαναλάβετε. Ποιο ήτανε? Για τη Frontex στην Ελλάδα ρωτήσατε για κάποιο hot spot στην Ελλάδα, κέντρο καταγραφής. Το ρόλο της Frontex στην Ελλάδα, λέει ο Πρόεδρος. Ε, I'm not Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα πάρα πολύ καλά το πνεύμα της ερώτησης, αλλά ποια είναι η άποψή μου για το ρόλο της Frontex με αυτή τη νέα ιδέα των κέντρων καταγραφής hot spots και την βοήθεια για την ταυτοποίηση και την καταγραφή στα σύνορα, κυρίως στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Υποθέτω ότι θα βοηθήσουν και στο θέμα της επανεγκατάστασης των προσφύγων, των ανθρώπων αυτών. It's true, Είναι γεγονός ότι φαίνεται απαραίτητη η παρουσία τους εκεί όταν είναι τέτοιες οι δυσκολίες σε ένα κράτος μέλος και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια κρίση. Καμιά φορά τίνουμε να κατηγορούμε ε, τις ε, παραμεθόριες χώρες ενώ το πρόβλημα είναι κοινό. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της Frontex στη μελέτη μας και αυτό που, πώς να το πω, διαπιστώσαμε από την ανάλυση και την έρευνά μας είναι το εξής. Εμείς επικεντρωθήκαμε στις σχέσεις με τρίτες χώρες, της σχέσεις της Frontex. Και εκεί είναι πάρα πολύ θολό το τοπίο και συγκεχημένη η εικόνα του τι γίνεται. Μπορεί να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια η διαφάνεια, ας πούμε, συνεργασίες και συμφωνίες με τρίτες χώρες για τη, της Frontex. Είναι εμπιστευτικά στοιχεία, το ξέρετε αυτά. Ε, η Frontex έχει αυτή την πολιτική της παθητικής δημοσίευσης. Δηλαδή οι ίδιοι δεν δημοσιεύουν τίποτα. Τα δημοσιεύουν κάποιοι άλλοι τα στοιχεία αυτά. Και βέβαια πάντα ανταποκρίνεται στα αιτήματα και στα ερωτήματα δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο αυτών των συνεννοήσεων και των συμφωνιών, αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις σχέσεις Frontex με τρίτες χώρες. Δεν ξέρουμε τι κάνει ακριβώς στα πλαίσια των συμφωνιών που έχει και των συμφωνιών που έχουν τα κράτη-μέλη με τις τρίτες χώρες. Δεν τα έχουμε αυτά τα στοιχεία γιατί δεν είναι δημόσια. Η Frontex κανονίζει γενικώς είναι διοικητικές συμφωνίες, δεν είναι συνθήκες διεθνείς ούτε συμβάσεις. Ε, θεσπίζουν ένα τρόπο θεσμικής συνεργασίας. Αλλά το πιο επίμαχο, κατά την άποψή μας, είναι κατά τη διάρκεια των περιπολιών ε, σε χωρικά ύδατα. Δεν μπορούν λοιπόν οι συμφωνίες εργασίας της Frontex να χρησιμοποιηθούν ως νομική βάση για τέτοιες κοινέ περιπολίες. Δεν έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα η Frontex για να εκτελεί ελέγχους στα σύνορα, να φυλάσει σύνορα. Λοιπόν, συνεννοήσεις κάνει και κάποιες συμφωνίες τέτοιου είδους συνεργασίας με τις χώρες οι οποίες δεν είναι δημόσιες επαναλαμβάνω και δεν κοινοποιούνται. Φαντάζομαι ε, ότι πρόκειται κυρίως για θέματα ασφαλείας. Τρίτες χώρες που συνεργάζονται με τη Frontex δεν θέλουν να δημοσιεύονται αυτά τα στοιχεία. Ούτε τα κράτη-μέλη. Γιατί τίθενται θέματα ασφαλείας. Ούτε μπορούν να ανακοινώνουν ότι σήμερα περιπολούμε στο τάδε σημείο και σήμερα επιχειρούμε στο δίνα σημείο. Όμως χρειάζεται πάρα πολύ περισσότερη διαφάνεια στα πεπραγμένα της Frontex και στις δραστηριότητές της όταν προσπαθεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη συνεργαζόμενοι με τρίτες χώρες. Και εμείς δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ανάληψη των ευθυνών τους. Η Frontex διαχειρίζεται εκεί ε, κάποιες επιχειρήσεις, αλλά το κράτος μέλος έχει την ευθύνη. Δεν ξέρω αν σας απάντησα, αν σας κάλυψα για αυτό που με ρωτήσατε. And, uh, well, I think it was not, Δεν ξέρω, αυτό ρωτήσατε. Remark, but thank you very much. Uh, ήταν μάλλον σχόλιο, δεν ήταν ακριβώς ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πιο προβληματικό θα είναι σίγουρα η πολιτική των επιστροφών. Right, uh, Uh, δεν ξέρω αν ήταν έκπληξη. Πάντως βλέπουμε τις τελευταίες εξελίξεις μετά ε, τη σύνοδο της Βαλέτα το πρόγραμμα δράσης με την Τουρκία. Επανέρχεται το θέμα των επιστροφών και των ασφαλών επιστροφών και δεν ξέρω ε, αν θα εφαρμόζεται το ΓΑΜ και σε ισορροπημένο, αλλά Ακόμα και η συμφωνία στα χαρτιά έχει ε, αθετηθεί όταν πρόκειται για την ασφάλεια, για την προσφυγική κρίση. Ε, η επιστροφή είναι το θέμα. Ευχαριστώ. Και μόνη η απάντηση. Ευχαριστώ, δόκτωρ Αντράντε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και μας παρουσιάσετε. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, και σας για τις ερωτήσεις σας. Και προχωρούμε. Στο σημείο 12 πάμε τώρα. Ο συνάδελφος Ζεράρντε Πρέ δυστυχώς κολλείεται σήμερα και απουσιάζει και το θέμα του θα αναβληθεί. Uh, uh, Ζητώ συγγνώμη και πάλι από τους συναδέλφους που παρέμειναν και περίμεναν το θέμα αυτό στο σημείο 13. Ο κύριος Ντεγιόνκ είναι καθοδόν και καθώς τον περιμένουμε θα μπορούσατε ίσως ξέρω εγώ, να ψυχαγωγηθείτε. Και μπορώ να σας πω, για να κερδίσω ένα μικρό στίχημα που έχω βάλει 2 ευρώ με τη γραμματεία, ότι θα προλάβαινα να τα πω αυτά πριν έρθει ο κύριος Δε Γιόγκ. Πάμε στο 13, μάλλον φαίνεται να το κερδίζω το σύστημα. Πάμε στο 14, συγγνώμη, 13 του κυρίου Δε Γιόγκ. Ε, εδώ βλέπω ότι είμαι εγώ εισηγητή και το ψιλογνωρίζω το θέμα. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειε κυκλοφορία οχημάτων ΑΚΟ στη Λετωνία, για όσους δεν γνωρίζετε τι είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με τη Συμφωνία Πριμ. Είναι το 14, παρουσίαση σχεδίου έκθεση από τον υποφαινόμενο στις 23 Νοεμβρίου αποφάσισαν οι συντονιστές, σας ευχαριστώ πολύ δόκτωρ, αποφάσισαν οι συντονιστές να, ε, να θέσουν στην ΚΟΕ την έκθεση και η ΚΟΕ μου είπε να τον αλάβω εγώ ε, με την ε, θεσμική μου ιδιότητα και κατ' εξαίρεση το ανέλαβα γιατί υπήρχε θέμα προθεσμιών. Θα το συζητήσουν αυτό όμως οι συντονιστές στην επόμενη συνεδρίαση. Ωραία. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών Ε, χαιρόμαστε όλοι για την ε, καλύτερη εφαρμογή της λεγόμενης απόφασης ΠΡΟΥΜ για την αυτόματη αλλαγή στοιχείων ε, ως προς την καταχώρηση οχημάτων από την Λετωνία. Ξέρετε ότι πολλές χώρες δεν ανταλλάσσουν τα στοιχεία που έχουν για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, ενώ αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο της Συμφωνίας ΠΡΟΥΜ και πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Συμφώνησαν λοιπόν οι συντονιστές να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου, γι' αυτό όλα τα αναλαμβάνω εγώ με τη θεσμική μου ιδιότητα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών μόνο στα αγγλικά, 14 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Monday. Είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται. Στη Λίμπε θα ψηφίσουμε 21 Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια 2 Φεβρουαρίου. Ελπίζω να μην θέλει κανείς να πει τίποτα φοβερά πράγματα. Είστε όλοι εντάξει, χαρούμενοι και ευτυχείς. Καλά, ευτυχείς. τώρα δεν είναι εύστοχο. Σχόλια. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. I'm two euros richer. Ορίστε, πλούτησα κατά δύο ευρώ. Ποιος τη χάρη μου. Uh, λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στο 13 που είναι το θέμα του κυρίου Ντεγιόγκ. Νομική συνδρομή για υπόπτου ή κατηγορουμένου που στερούνται τη ελευθερία του και τη νομική συνδρομή σε διαδικασίε εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη. Περιμένουμε ανυπόμονη τον κύριο Ντεγιόγκ. Από στιγμή σε στιγμή. Μόλις έρθει εννοείται ότι θα τον καταχειροκροτήσουμε, ούτε rock star να ήταν. Ζητώ συγγνώμη που σας υποβάλλω σε αυτή τη δοκιμασία. Τι άλλο να πούμε. Ήρθε, ήρθε, ήρθε. I'm sorry, Mr. De Jong, my uh, a mixture of tiredness, a couple of painkillers and uh, various other things. Okay. Μάλιστα. Εντάξει, ε, είχα την ευκαιρία να διεκπαιρεώσω τη δική μου έκθεση και ας έχει μείνει μόνο το δικό σας θέμα για σήμερα. Θα σας έλεγα ακόμα και την, τα διάφορα και τις προσεχείς συνεδριάσεις, αλλά εντάξει έχουμε μερικά σημεία ακόμα μέχρι τότε. Περιμένω λίγο να καθίσετε και να τακτοποιηθείτε κύριε Ντεγιόγκ για να ετοιμαστείτε να τα πείτε. Λοιπόν, νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους που στερούνται της ελευθερίας τους και τη νομική συνδρομή για διαδικασία εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Είναι παρουσίαση του θέματος της πρόοδου των τριμερών διαπραγματεύσεων στην Επιτροπή. Άλλο σημαντικό θέμα θα μας πει τώρα ο κύριος De Jong τι γίνεται. Τελευταίος τριμερής διάλογος έγινε στις 18 Νοεμβρίου και να ακούσουμε πραγματικά που βρίσκεται το θέμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Ντεγιόγκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Την περασμένη φορά ήμουν πολύ αρνητικός, τώρα είμαι λιγότερο αρνητικός. Είμαι αρνητικός σκέτο, πράγμα που συνιστά βελτίωση. Δεν είναι μόνο άσχημα τα νέα, ε, αφού συναντηθήκαμε με τους σκιώδεις ηγητές, συνεδρίασα με τον Υπουργό Δικαιοσύνη των Κάτω Χωρών και συμφωνήσαμε στην Ολλανδική Προεδρία να δοθεί σοβαρά προσοχή σε αυτό το θέμα με στόχο να επιτευχθούν και αποτελέσματα. Θετικά ελπίζουμε. Η αρνητικά θα δείξει Πάντως ε, θα δούμε, θα δούμε ποια θα είναι η έκβαση. Πάντως ε, πρόθεση έχουν και οι δύο πλευρές να γίνει μεγάλη πρόοδο στο επόμενο εξάμεινο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε ούτε ημερομηνία ούτε ώρα για φέτος ακόμα οπότε ε, δεν πρόκειται η Λουξεμβουργιανή Προεδρία να κάνει άλλους ε, τριμερείς διαλόγους. Αρχές Ιανουαρίου, το πολύ μέσα Ιανουαρίου θα είναι ο επόμενος τριμερείς διάλογος υπό Ολλανδική Προεδρία πλέον. Με το καλό. Ως γενική προσέγγιση Πρέπει να πω ότι και με τους σκιώδεις ηγητές και με την Προεδρία του Συμβουλίου συμφωνήσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε είναι να επικεντρωθούμε στο άρθρο που έχει να κάνει ε, με καταζητούμενους ε, με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ε, αλλού υπάρχει πρόβλημα αναλογικότητας κτλ. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσέγγισης. Μπορούμε να συζητήσουμε αρκετά πράγματα ε, που μπορούν γενικά να εφαρμόζονται και αλλού, αν συμφωνήσουμε ότι σε απότερο στάδιο θα εφαρμοστούν και σε άλλες περιπτώσεις. Στον τριμερή διάλογο ξεκαθαρίσαμε ότι αν ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση δεν σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα κάνει πίσω, ούτε πρόκειται να υποχωρήσει σε τίποτα από τη θέση του ως προς το πεδίο εφαρμογής. Δηλαδή υποχωρήσεις και παραχωρήσεις δεν κάνουμε, μην νομίζει κανείς, ε, απλώς ε, αρχίζουμε ε, τα γνωστά στους τριμερείς διαλόγους, ε, κάποια κείμενα να γράψουμε για να συζητούμε από αυτόν. Επιπλέον, και αυτό ήταν μέτρο ε, οικοδόμηση εμπιστοσύνης, πιστεύω ότι θα είναι προς όφελος και του Κοινοβουλίου και συμφωνήσαμε αν το εγκρίνουν τη Δευτέρα βέβαια οι συντονιστές, δεν θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να κάνει μια μελέτη αντικτύπου για τις αλλαγές που προτείνουμε σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το συγκρίνουμε δηλαδή με το τελικό αποτέλεσμα, σε περίπτωση που εγκριθεί η δική μας προσέγγιση και πρόταση σε διάφορους τομείς. Εντάξει, μπορεί κανείς να σκέφτεται το κόστος και τις διοικητικές δαπάνες, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις οικονομίες. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί όταν ε, δίνεις νομική συνδρομή αρρωγή σε κάποιον στην αρχή μιας ε, διαδικασίας μπορεί τελικά να εξοικονομήσεις χρήματα ε, εκ των υστέρων. Ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε με τους και είναι και συμφωνήσαμε γενικά και θα πρέπει να το επικυρώσουν οι συντονιστές. Ζητήσαμε νομική ε, βοήθεια, συμβουλή, άτυπη, όχι, όχι επίσημη γιατί αυτό παίρνει πολύ χρόνο, αλλά να μας δώσουν κάποιες άτυπες απαντήσεις ως προς το πεδίο εφαρμογή πρώτα της οδηγίας για την ε, το δικαίωμα για πρόσβαση σε νομική συνδρομή σε δικηγόρο, αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28, διότι η Προεδρία λέει σε έγγραφο του Συμβουλίου ότι σύμφωνα με εκείνους, με βάση αυτές τις αιτιολογικές σκέψεις δεν υπάρχει υποχρέωση να δίνεται δικηγόρος ή νομική συνδρομή όταν δεν υπάρχει στέρηση ελευθερίας, όταν δεν είναι δηλαδή κρατούμενος ο άλλος. Ε, θα πρέπει να το κοιτάξει αυτό η νομική υπηρεσία. Εγώ δεν συμφωνώ με την Προεδρία δεν έχουμε τέτοια θέση εμείς, ούτε τέτοια ερμηνεία. Αλλά θέλω να το μελετήσουμε, να μας βοηθήσει η νομική υπηρεσία για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Επίσης, ένα άλλο που είναι γενικότερο σημείο και για να δείξουμε επίσης ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που από όλο το πακέτο και τον οδικό χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα ε, ε, διαφωνούμε για όλα εκτός από τη νομική συνδρομή. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν η νομική υπηρεσία να εξετάσει και πάλι άτυπα, όχι με την επίσημη διαδικασία, ποια θα ήταν η συνέπεια εάν, αν, για παράδειγμα, ένας καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης πει μου στέρισαν την νομική συνδρομή Και το γεγονό ότι υπάρχουν τώρα ευρωπαϊκά πρότυπα για νομική διαρρογή και συνήγορο και δεν μου έχουν δώσει δικηγόρο, αλλά εγώ δεν μπορώ να ε, ε, αντιταχθώ στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα τέτοιο πλαίσιο, οπότε έχει ενδιαφέρον αυτή η σχέση και ε, έχει ενδιαφέρον για ποιο λόγο. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν τη θέλουν καθόλου αυτή την οδηγία και θέλουν να την ξεφορτωθούν. Γι' αυτό θα ήταν από πλευρά μα ένα επιχείρημα που θα πει ανεξαρτήτως της μορφής που θα πάρει αυτό κάποια νομική αρρωγή θα πρέπει να δεχθείτε. Ελπίζω οι συντονιστές να υποστηρίξουν τη δική μας προσέγγιση. Έχουμε και τη μελέτη αντικτύπου. Φυσικά μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου μου είπανε. Νομίζω είναι καλή αυτή η συγκυρία και ο χρονισμός και θα μπορούσε η Γενομική Υπηρεσία να μας έχει απαντήσει και νωρίτερα σε λίγες εβδομάδες, δηλαδή κάπου στο Γενάρη. Ας το συζητήσουμε με την Προεδρία και εγώ προσβλέπω, ελπίζω σε επικοδομητικές συζητήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεγιόγκ. Εγώ το έχω παρακολουθήσει λίγο αυτό το θέμα και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και σας εύχομαι κάθε επιτυχία με την Ολλανδική Προεδρία. Δεν είναι τεχνικά δύσκολο, αλλά πολιτικά ε, ε, μπορεί να υπάρχουν ε, ε, αντιστάσεις, γιατί έχουν γίνει πολλές περικοπές σε αυτό τον κλάδο εδώ χρειάζεται χρηματοδότηση για να τηρηθούν κάποιες διαδικασίες οι οποίες καταραίουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και το όλο το σχέ με πολλούς τρόπους. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις αρχές του 2016. Η κυρία Τσινίτσελ, μια συνάδελφος που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, Κατρίνα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους της κυρία Σίπελ, οπότε θα τα προσπαθήσω στα αγγλικά. Η Birgit ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ε, έχει το τακτικό του συνέδριο στο Βερολίνο όμως μου ζητά να εκφράσω την πλήρη στήριξή της προς την προσέγγιση του εισηγητή. Η μελέτη επιπτώσεων των βασικών μας τροπολογιών καθώς και το να ζητήσουμε από την νομική μας υπηρεσία νομικές διευκρινήσεις είναι κάτι που θα μας επιτρέψει να έχουμε σταθερότερα επιχειρήματα για να προβάλλουμε τη θέση μας ασχέτως των ε, πολύ αδιάλεκτων ε, απόψεων του Συμβουλίου εδώ, δεν θα πρέπει να ενδώσουμε και να εγκαταλείψουμε τη δέσμευσή μας για δίκαιη εκδίκαση των υποθέσεων οποιοδήποτε υπόπτου ή κατηγορουμένου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν. Όχι. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Τεκιόγκ. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλό κουράγιο με την Ολλανδική Προεδρία που είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ δραστήρια. Συναντήθηκαμε με τον πρέσβη και με υπαλλήλους και του θέσαμε υπόψη αυτό το σημαντικό θέμα μεταξύ άλλων ε, και τους έχουμε επισημάνει ότι μας ενδιαφέρει πολύ. Λοιπόν, ας το προωθήσουμε. Λοιπόν, συνάδελφοι, πριν φύγετε, αφού διεκπαιρέωσα και τα δικά μου θέματα πάρα πολύ γρήγορα, στο 16 είναι προσεχή συνεδριάσεις, 17 ε, Δεκεμβρίου ημέρα 5η, 9.30 στο Στρασβούργο. Είδατε τι κατάφερα. Κατάφερα να μου εγκρίνουν συνεδρίαση της Επιτροπής στο Στρασβούργο. Που έτσι κι αλλιώς στο Στρασβούργο είδα προβλήματα πολλά. 9.30 με 10 και μετά 21 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες και 22 Δεκεμβρίου επίσης στις Βρυξέλλες. Διάφορα δεν έχουμε. Έχει κανείς κανένα διάφορο. Όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι για τη σημερινή σας ε, προσέλευση και παραμονή. Το εκτιμώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα για όσους παρέμειναν καθόλου όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.